Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη να καθίσετε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση. Υπάρχει κάποιος του ΕΛΚ, υπάρχει κανείς του ΕΛΚ στην αίθουσα. Right. Ας τα ψηφίσουμε όλα μαζί με τη μία, ορίστε, πάμε. θα αναφερθώ στο θέμα των ενδιαφέρων των διαφόρων εκχωρημένων πράξεων. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αν έρχεται, α, αν έρχεται διαδικαστικό, η Αρλίν θα ασχοληθεί με το θέμα. Όπως είμαι σίγουροι ότι γνωρίζουν τα μέλη, πρόκειται περί γνωμοδοτήσεως που υποβάλλεται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων όσον αφορά τις εκχωρισμένες πράξεις, ανατεθήσεις πράξεις, που είναι κάτι που αφορά την διαδικασία επιτροπολογίας, πώς αλλιώς να το πούμε, λήψη καλύτερης έκφρασης και έχουμε και κάποιες προταθήσεις ε, τροπολογίες και έχουμε και κάποιες συμβαστικές τροπολογίες όπου, με τις οποίες οι περισσότεροι συμφωνούν. Αν καταφέρω να τις βρω βέβαια τις τροπολογίες. Είναι στον κατάλογο ψηφοφοριών. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες που έχουμε αφορούν την τροπολογία 6. Έχουμε συμπλήρωση στο τέλος, υπενθυμίζοντας ότι σε όλους τους τομείς η βασική πράξη οδηγίε, οι βασικέ πράξει, οδηγίε κλπ. θα πρέπει ρητά να αναφέρονται στο στόχο περιεχόμενο, πεδίο και διάρκεια τη εκχωρηθή σα ε, πράξη και τι προποθέσει υπό τι οποίε γίνεται αυτή η εκχώρηση για να διευκρινιστεί η διαδικασία, η επόμενη προφορική τροπολογία είναι, αφορά την παράγραφο 4 και τελική πρόταση για την αλόγω παράγραφο λέει «Καθορίζω ότι οι συνθήκες δεν καθορίζουν οδήποτε απέτηση για νομοθετικές αποφάσεις επί πράξεων να συμπεριλάβουν γραπτές εξηγήσει για θέτηση ε, ακύρωση εκτός από τις γενικές υποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 296 του Ευρωπαϊκή Ενώσεω, που είναι κάτι που ισχύει για τι νομικέ πράξεις, συνθήκη ΕΟΚ. και νομίζω ότι συμφωνήσαμε επ' αυτών των δύο προφορικών τροπολογιών. Τα υπόλοιπα θα υποβληθούν συλλογικά. Δεν ξέρω αν κανείς από τους παρόντες επιθυμεί να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις ή να συζητήσει αυτές τις τροπολογίες. Υπάρχει κανείς που να γνέφει, όχι. Οπότε εάν υπάρχει μια γενική συμφωνία από αυτόν, διότι το συζητήσαμε επί μακρόν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω email, θα ήταν καλό να γίνει μια ψηφοφορία, να τις ψηφίσουμε ομαδικά όταν φτάσουμε στην ψηφοφορία και η γραμματεία πιθανότατα θα προσπαθήσει να τις επαφεί με τους ε, συντονιστές που λείπουν πριν την ψηφοφορία επί του θέματος. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να πάμε σε πιο ενδιαφέροντα θέματα παρόλο που θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι κάτι αμεληταίο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξέταση του σχεδίου εκθέσεως σχετικά με το CRD3 και θα δώσω το λόγο στην Αλήν Μακάθη το λόγο για την ε, παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχω τη δυνατότητα, να είχα τη δυνατότητα το συζητήσαμε δύο φορές θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε κάποιες από τις ανησυχίες ή κάποιες από τις ιδέες που έθεσαν κάποιοι σε αυτή την συζήτηση και βέβαια έχοντας υποβάλει την έκθεση μπορώ να συζητήσω και με τα μέλη διμερός και με τους κοιόδης να δούμε τι τροπολογίες που υποβληθούν. Μα η βασική ιδέα είναι η ίδια. Αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, αυτή την οδηγία, διότι οι τράπεζες είχαν πολύ λίγα κεφάλαια και ο κίνδυνο μοντέλων των τραπεζών έβρισκαν ε, ότι χρειαζόταν όλο και λιγότερα κεφάλαια για τι εμπορικέ διαδικασίε και πέρα από αυτό ε, υπήρχε και η κουλτούρα των πόνου των αρχιπρόθεσμων και με την έλλειψη κεφαλαίων που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό όσον αφορά την οικονομική κρίση είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εξετάζοντα λοιπόν την προσέγγιση που θα ήθελα να ακολουθήσω όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση πρέπει να πω ότι η πρώτη μου ευθύνη ήταν ε, νομοθετική. Είναι νομοθετική σε αυτή την Επιτροπή. Θέλω να δω ποια είναι τα συμφέροντα των, ε, του κοινού των φορολογουμένων και συζητήσαμε εκτενώ αυτά τα θέματα μέσω του τύπου, μέσω των μέσων ενημέρωση. Επίση, είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και στι πρώτερε δύο συζητήσει, ανταλλαγέ απόψεων και νομίζω ότι όλοι μα συμφωνούμε ότι ο στόχο είναι ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ισχυρότερο, σταθερότερο τραπεζικό σύστημα που δεν χρειάζεται να, να το γλιτώσουν οι φορολογούμενοι, ότι οι πολιτικέ αμοιβών δεν θα πρέπει να θαρρύνουν υπερβολική ανάληψη κινδύνων και γι' αυτό αυτό που κάνουμε στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώση να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε ε, κανόνες στεναρούς αλλά δίκαιους. Ε, μπορούμε να αναθεωρούμε μακροπρόθεσμα την οδηγία αλλά δεν θέλουμε να έχουμε έναν ε, μοναδικό ενιαίο υπερφόρο και μέτρα που καλύπτουν και ανά θέλουμε να προσέξουμε τι θα θεσπίσουμε για πιο μακροπροθεσμε λύσει. Και γι' αυτό το λόγο οι τροπολογίε μου ακολουθούν ε, τι αρχέ ε, τη αρχή για την χρηματοσυντική σταθερότητα που συμφώνησαν οι G20. Χρειαζόμαστε μια γενική προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το τομέα. Αυτέ οι πολιτικέ που θετούθε από του G20 είχαν σαν στόχο να σταματήσουν την υπερβολική ανάληψη κινδύνων να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αποδυναμώσουμε τα χρηματοστικά ιδρύματα και να υποστηρίξουμε τη σωστή διαχείριση των κινδύνων. Και αυτό που έκανα και νομίζω ότι και τα μέλη που θέλουν να το εξετάσουν λεπτομερέστερα το θέμα θα δουν ότι έχω συμπεριλάβει ουσιαστικά αυτά που είχαμε στι συστάσει μα, στι προτάσει σχετικέ και τα συμπεριλάβαμε σε νομοθετική μορφή για κατορισμό. Θα συνταχθούν διαφορετικά στην τελική μορφή. Διότι δεν μπορεί να συντάξει ένα νομοθέτημα με αοριστολογίε και αόριστε συστάσει. Θα δείτε λοιπόν ότι είναι λεπτομερέστερε και πώ έχω συντάξει αυτέ τι προτάσει και όπω είπα μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές εκεί που υπάρχουν ασάφειες, εκεί που θα πρέπει να δώσουμε κάποιες αποσαφηνίσεις Θα ήθελα να επιθυμίσω στους συναδέλφους ε, ποια είναι η αρχή αυτού που συζητούμε και γι' αυτό συνέταξα και τις, αυτές τις προτάσεις. Ότι τα μπόνους θα πρέπει να είναι αμοιβή για σωστή μακροπρόθεσμη επίδοση και της εταιρεία και του ατόμου. Θα πρέπει να είναι ανάλογα αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να αντικατοπίζουμε στι τροπολογίε που παβάλλουμε και δεν θα πρέπει να είναι εγγυημένα αυτά τα μπόνου. Λοιπόν, εφαρμόζοντα αυτέ τι αρχέ στην ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία, εξακολουθώ να λέω ότι είναι ευθύνη των εταιριών να αποφασίζουν ποια είναι η αμοιβή οι αμοιβέ που δίνουν και είναι ευθύνη των εθνικών εποπτικών αρχών να εξασφαλίσουν ότι αυτέ οι πολιτικέ ευθυγραμμίζονται με τι διάφορε πολιτικέ, αλλά όπω σα είπα, έλαβα υπόψη τις αρχές από το αρχικό κείμενο με κάποιες μικροαλλαγές που επίσης σας εξηγώ. Αλλά να κάνω μια επισκόπηση τώρα των βασικών αρχών που έχουν συμπεριληφθεί στην οδηγία και κάποιε αυτέ τι αρχέ ήδη έχουν συμπεριληφθεί από το Συμβούλιο στη, στο έγγραφο εργασία του Συμβουλίου. Τα μπόνου θα πρέπει να δίδονται επί τη βάση μακροπροθέσμων επιδόσεων και να μην υπάρχει εγγύηση, να μην υπάρχουν χρυσά λεξίπτωτα αν υπάρχει αποτυχία. Θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα των εταιριών, αυτή είναι η προτεραιότητα. Γι' αυτό οι πληρωμέ των μπόνου των εταιριών δεν θα πρέπει να περιορίζουν τη δυνατότητα που έχουν να ισχυροποιούν το κεφάλαιό του, την κεφαλαιοκή του βάση και 50% τουλάχιστον των μπόνου θα πρέπει να καταβάλλεται σε, μερίδια, σε μετοχέ. Και αυτό που έκανα στην πρόταση είναι να κοιτάξουμε τη σύσταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι αμοιβέ του 2009 που λέει ότι αυτέ οι συμμετοχέ θα πρέπει να κρατούνται τουλάχιστον για τρία χρόνια και θα δείτε, συνάδελφοι, ότι πολλέ τράπεζε τώρα έχουν εισάγει αυτό το δελογικό κώδικα, τον έχουν επιβάλει στον εαυτό του όσον αφορά ε, την κράτηση των μετοχών για μία τριετία. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να αναβληθούν τα μπόνους κατά αναλογία με τον επιχειρηματικό κύκλο, με τον κύκλο εργασιών. Αυτό είναι κάτι με τον κύκλο, τη διάρκεια, τη χρονική των εργασιών. Οι εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να, το εξετάσουν. Και αυτό το κομμάτι που αναβάλλεται θα πρέπει να ανακαλείται αν υπάρχουν επιδόσει κατώτερε των αναμενόμενου. 40% του μπόνους, 60% για πολύ μεγάλα μπόνους θα πρέπει να αναβάλλεται η καταβολή του και η περίοδο αναβολή θα πρέπει να είναι μικρότερη από τα τρία χρόνια. Οι εταιρείε θα πρέπει να έχουν μια επιτροπή αμοιβών που θα αναθεωρεί και θα εξετάζει τι πολιτικέ που ακολουθούνται και προτείνω. Ο πρόεδρο και η πλειοψηφία των μελών τη επιτροπή. θα πρέπει να μην ανήκουν στο διοικητικό στελέχη, να μην είναι εκτελεστικοί διευθυντέ και θα το εξετάσω αυτό διότι θα δείτε ότι είπα, ανακοίνωσαν στο δικό τους νομοσχέδιο ότι θέλουν 100% των μελών να μην ανήκουν στη, να μην είναι διευθυντικά στελέχη, εκτελεστικοί διευθυντές. Οι επιχειρήσει θα πρέπει να αποκαλύπτουν δημοσία τι πληροφορίε σχετικά με τι αμοιβέ που δίνουν και τι πληρωμέ και αυτό είναι περιγραφή τη αρχική πρόταση και προσέθεσα κάποια πράγματα εγώ ότι αυτές τις πληροφορίες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πληρωμές από τη μονάδα της επιχείρησης να καταλάβουμε ποιες δραστηριότητες, ποια μπόνους ε, συνδέονται ποιες δραστηριότητες. Δώσω πρακτικό παράδειγμα. Αυτή την εβδομάδα Μεγάλη Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε ότι πλήρωσε 2,2 δις τον πόνους για για δραστηριότητε απροσδιορίστου κινδύνου τη εταιρεία. Η άποψή μου πρέπει να ξέρουμε ποιε δραστηριότητε είναι αυτέ. Ποια επιχειρηματική δραστηριότητα δέχτηκε τα 2,2 ε, δισεκατομμύρια σε Σύμφωνα με τη σύσταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 204-943 που αναφέρεται στην καλύτερη διακυβέρνηση, προτείνω αυτή η πληροφορία να δημοσιεύεται σε ατομικό επίπεδο για του ε, διευθυντέ των τραπεζών και θα ήθελα να τονίσω δύο τομεί, όπου εκεί ενίσχυσα κάπως το κείμενο εν συγκρίση με το αρχικό και τις προτάσεις. Η αρχική πρόταση έλεγε ότι προέβλεπε ειδικά μέτρα για τις τράπεζες που χρειάζονται βοήθεια και είδαμε ότι πολλές χώρες έκαναν αυτά, ακούσαμε την προσέγγιση σε περίπτωση των ε, εταιριών που είχαν πρόβλημα και υπήρχε αυστηρό έλεγχο στη ΣΥΠΑ όσον αφορά τι αμοιβέ των διευθυντών. Και πρότεινα μια τροπολογία, τροπολογία 53, κάποιε πτυχέ αιρεσιμότητα και πριν παρεξηγηθώ για αυτά που έκανα, δεν είπα ότι θα πρέπει να επαγορευτούν τα μπόνους για τις τράπεζες που έχουν βοηθηθεί, αλλά τα μπόνους θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, υπάρχουν κάποιοι όροι. Δηλαδή η εταιρεία ή η τράπεζα θα πρέπει να οικοδομεί την κεφαλιακή βάση της εταιρεία και να αποπληρώνει τους φορολογουμένους. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση και μετά να πληρώνται τα μπόνους. Αυτό είναι μόνο σε, είναι εξαιρετικό μέτρο, προσωρινό μέτρο για ε, τράπεζε που στηρίζονται από τα χρήματα του φορολογωμένου. Θέλουμε να βελτιώσουμε σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των εταιριών. Δεν θέλει κανεί από εμά και το κοινό δεν συμφωνεί. Τράπεζε οι οποίοι ε, είχαν απώλειε και του βοήθησε φορολογούμενο, το πρώτο που κάνουν είναι να πληρώσουν εμπόνου σε εταιρείε. Αυτό είναι, θα είναι κατά τη αρχή του αρχικού κειμένου, διότι θα βραβεύεται η αποτυχία. Άρα είναι μια παραβίαση των αρχών του αρχικού κειμένου του FSB και κάτι άλλο που πρόσθεσα στην, προ... αρχική πρόταση ήταν ότι τα μπόνους θα πρέπει να είναι αναλογικά με τους μισθούς. Συνάδελφοι, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς να μην συμφωνείτε με την πρόταση που υπέβαλα, όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο να καθορίσουμε τι σημαίνει αυτή η αναλογικότητα, αυτό όρο. Δεν αρκεί να λέμε ότι πρέπει να είναι κάτι αναλογικό. Αυτό που προσπάθησα να κάνω εδώ είναι να πάρω το μοντέλο το Ολλανδικό. Οι Ολλανδοί έχουν εφαρμόσει μέσω τραπεζικού του κώδικα μια απέτηση τα μπόνου να μην ξεπερνάνε το μισθό. Ε, πιστεύω ότι αυτό είναι σαφό μέτρο αναλογικότητα ή ένα τρόπο προσμέτρηση αναλογικότητα. Σε οποιοδήποτε μέρο του κοινού θα μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Οπότε έχουμε τροπολογία 55, από εκεί προτείνω ότι η συνολική μεταβλητή αμοιβή να μην είναι πάνω το 50% από τη συνολική αμοιβή ενό ατόμου σε ένα χρόνο. Όπω είπα, μπορούμε να βρούμε και άλλου τρόπου για να καθορίσουμε ή να θέσουμε ε, πιο ουσιαστικά το θέμα του τι είναι αναλογικό. Είναι πολύ δύσκολο, συνάδελφοι, να δούμε πώς θα μπορούσε να υπάρχει συνέπεια με την αρχική απέτηση του αρχικού κειμένου, FSB, και κατά πόσο θα ήταν δυνατόν να μην πληρώνονται μπόνους και οι γενικές δομές αμοιβών να μην ενθαρρύνουν τον υπερβολικό κίνδυνο. Είναι τεράστια πλειοψηφία το, το, το, το, τεράστιο, το 90% ε, των εισοδημάτων κάποιου να προέρχονται από τα ε, μπόνους αν εξαρτάται κανεί κατά πολύ από τα μπόνου, δεν πρέπει να σπάσουμε τη σύνδεση μεταξύ αμοιβή μεσομπόνου και αναλήψεω εξαιρετικού κινδύνου. Υπάρχει ένα τρόπο αυτό να πετύχουμε μια ισορροπία, αλλά είμαι ανοιχτή και σε κάποιε προτάσει. Έχω προτείνει οι εθνικέ εποπτικέ αρχέ θα πρέπει να βαθμολογήσουν τι αμοιβέ και τα μπόνου ε, σε όλε τι εταιρείε. Έχω προτείνει ότι οι εθνικέ εποπτικέ αρχέ να βαθμολογούν να βλέπονται ποιε είναι οι πολιτικέ αμοιβών και μπόνους στα κάτι μέλη στι διάφορε εταιρείε. Αλλά αυτό που έκανα επίση να προσθέσω και μία απέτηση ότι αυτέ οι πληροφορίε θα πρέπει να διαβάζονται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, ούτω ώστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια προσπάθεια βαθμολόγηση, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώ αυτέ οι πολιτικέ προσπαθεια βαθμολογηση γιατι πιστευω οτι παρα πολυ σημαντικο να δουμε πω αυτε οι πολιτικε λειτουργουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Για να έχουμε αναφορέ και εκθέσει και όπου χρειάζεται να κάνουμε τι δέουσε προσαρμογέ. Διότι βεβαίω αυτή είναι μια πολύ καινούρια ε, πολιτική, ριζική απόκληση και ίσω είναι ένα τομέα στον οποίο χρειάζεται να κάνουμε προσαρμογέ στο μέλλον. Θέλουμε να κάνουμε προσαρμογέ. Τώρα πάω στο άλλο κομμάτι όσον αφορά τις κεφαλικές, ε, κεφαλουχικές απαιτήσεις πρέπει να είμαι ξεκάθαρη εδώ οι τροπολογίες μου που είναι πολύ λίγες, ελάχιστες τι προσπαθούν να κάνουν, να εφαρμόσουμε τις, τα διεθνώ συμπεφωνημένα, του κανόνε για κεφαλουχικέ απαιτήσει που προέρχονται από τη Βασιλεία. Οι τράπεζε ξέρω ότι σα χτύπαγαν τι πόρτε και εξέφραζαν ανησυχίε σχετικά με το θέμα και οι τράπεζε από ό,τι γνωρίζω είπαν ότι θα μοιραστούν μαζί μου ποιε είναι τροπολογίε που θα υποβάλουν για αυτό το κομμάτι τη εκθέσεω και ξέρω ότι οι τράπεζε είπαν ότι θα ήθελαν κάποια καθυστέρηση μέχρι το 2012 αλλά τώρα οι τράπεζες θέτουν και άλλες ανησυχίες περί του ποσού του κεφαλαίου που θα πρέπει να κρατήσουν, του υψού του κεφαλαίου και αν είναι πολύ ψηλό το κεφάλαιο, αυτό λένε ότι είναι πολύ ψηλό το κεφάλαιο και πρέπει να σταθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις της Βασιλείας. Δεν πρότεινα εγώ καμία καθυστέρηση στον αφορά το χρονοδιάγραμμα της Βασιλείας. Πιστεύω ότι για να το κάνουμε αυτό θα έπρεπε να έχουμε περισσότερα ανεξάρτητα στοιχεία αρνητικών συνεπειών στην πραγματική οικονομία σε σχέση με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμφώνησε να εφαρμόσει του υποφωνημένου διεθνεί αυτού κανόνε και δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα για καθυστέρηση ούτω ώστε να μην συμμορφωθούν και άλλε χώρε. Κατά πρώτον, εάν δεν προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε το χρονοδιάγραμμα, δεν θα μπορέσουμε να ζητήσουμε από άλλου να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει που ανελήφθησαν τον τελευταίο χρόνο, το 2009. Δεύτερον, ε, δεν πιστεύω ότι η εφαρμογή της, των κανόνων τη Βασιλεία ε, θέτει σε μειονεκτική θέση την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ανταγωνιστικά. Ε, δεν έχει νόημα να αυξήσουμε τι απαιτήσει μα αν τελικά χρησιμοποιούν περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων για να γλιτώσουμε τι τράπεζε. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί να διορθώσουν την υποτίμηση του κινδύνου ε, και όσον αφορά του τίτλου αξιόγραφα, αν δεν διορθωθεί αυτό, θα δημιουργηθούν νέα προβλήματα όσον αφορά τα ισοσύγια των τραπεζών και θα παραμείνουν τα ευάλωτα στοιχεία, δεν θα καλυφθούν επαρκώς, αναφισβήτητα θα πρέπει να προχωρήσουμε έγκαιρα όσον αφορά αυτά τα μέτρα ή ενδεχομένω να μην ξαναδιαπιστωθούν αποτυχίε τραπεζών. Τα στοιχεία ενεργητικού ε, θα πρέπει να προσέξουμε αν έχουν υποτιμηθούν τελικά τα δάνεια και τι κεφάλαιο συνδέεται με τα κεφάλαια που έχουν χορηγηθεί σε δανειοδότηση θα πρέπει να δούμε τι κίνδυνο για την εμπορική δραστηριότητα. Εάν φυλαμιστεί αυτό το κόστο, θα μειωθεί υπερβολικό τονισμό κάποιων στοιχείων και δεν θα είναι κάτι αντιπαραγωγικό ή την ιδιωτική δραστηριότητα. συμφωνήθηκαν το πρώτο εξάμεινο του 2009 αυτά στην Βασιλεία και οι τράπεζε είχαν πάνω από 18 μήνε συμμορφωθούν με την ημερομηνία εφαρμογή. Από όταν υπεγράφει αυτή η συμφωνία, οι τράπεζε ε, κάπω συμμαζεύτηκαν σε σχέση με το 2009 όσον αφορά τα μπόνους και τα μερίδια που δώσανε στους υπαλλήλους δείχνουν ότι μπορούν να συμμορφωθούν με τα τις εντολές της Βασιλείας υπάρχουν χρήματα εγώ αν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία μπορώ να κάνω προσαρμογές βάσει στοιχείων ότι αυτό, ε, τα μέτρα αυτά θα επηρέαζαν τη δανειοδοτική δυνατότητα που έχουν οι τράπεζε για να δανειοδοτούν την πραγματική οικονομία. Το τέλο 2010, αν το κρατήσουμε, εγώ προτείνω, σαν ημερομηνία εφαρμογή, θα επαγρυπνούμε όσον αφορά νέα στοιχεία, όσον αφορά τι μελέτε ποσοτική συνέπεια. Και αν δούμε ότι είναι σφαλμένε Εσφαλμένα τα πορίσματα τη εκθέσεω, τη προτάσεω μάλλον, θα κάνουμε εμεί τι δέουσε προσαρμογέ. Λοιπόν, οι πιο θεμελιώδεις αλλαγές του καθεστώτος Βασιλείας που θα μπουν στο CRD4, το Κοινοβούλιο ήδη ζήτησε μια πλήρη έκθεση από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά ε, το τέλος 2009, όσον αφορά το προηγούμενο πρόγραμμα εγώ ε, ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η έρευνα να τα πορίσματα αντιποβληθούν στο Κοινοβούλιο και να διαπραγματευτούμε στα πλαίσια τη Βασιλεία αν υπάρχει σαφή εντολή από πλευρά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οι θεμελιώδει αλλαγέ που προβλέπονται, όπω είναι το ποσοστό μόχλευση, φαινομένου μόχλευση κλπ. Η ε, δυναμική, ο δυναμικός εφοδιασμός και ελευθερία δεν είναι τεχνικές επιλογές, είναι θέματα τα οποία μπορεί να έχουν πολιτικό χαρακτήρα και γι' αυτό χρειάζεται έλεγχος του Κοινοβουλίου και είναι κάτι που έχω συμπεριλάβει σε διάφορες διατάξεις όσον αφορά τις εκχωρηθήσεις ανατεθήσεις πράξεις. Και το έκανα αυτά σύμφωνα με τη δουλειά που έκανε ο κύριος Σάντσες, τη δική του έκθεση, για την ε, οδηγία Omnibus 1. Οπότε έχουμε εκχωρηθεί ε, σε πράξει σε τρει τομεί. Αν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάποιε τεχνικέ προδιαγραφέ βάσει συμβουλή του CDEBA, θα πρέπει αυτέ να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με τι νέε εξουσίε που προβλέπονται εάν η Βασιλή συμφωνεί ότι θα πρέπει να υπάρχει κεφαλογική απέτηση ελάχιστη για τις ε, συναλλαγές, κάτι που συζητείτε, αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω εκχωρηθής σας εξουσίας, ανδεθής σας εξουσίας και πρότεινα ένα συμβιβασμό μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μέτρα που προτείνονται για πολύ περί... την πολύ περίπτωση διαδικασία αποτιτλοποίησης θα πρέπει να δείτε τη δέουσα προσοχή και θα πρέπει να δίνεται έγκριση από πλευρά υποπτικών αρχών σε αυτέ τι συναλλαγέ. Τα κράτη-μέλη είχαν αντιρρήσει. Πίστευαν ότι έτσι θα είναι πολύ επαχθή ο κανονισμό και ίσω να έχουν δίκιο σε αυτόν τον τομέα. Σαν συμβιβασμό, λοιπόν, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω την ανάγκη για τέτοιε διατάξει, κυρίω να δει κατά πόσο τα νέα μέτρα του CRD2 για την σωστή προσέγγιση είναι κάτι αποτελεσματικά και αν είναι αναγκαίο να υποβάλει μια πρόταση για συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια για πολύ περίπλοκη ε, αποτιτλοποίηση και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε και να συμφωνήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτά τα μέτρα Αυτά τα μέτρα πετυχαίνουν τη σωστή ισορροπία, πιστεύω, μεταξύ τη αναγκαία ευελιξία για να υπάρχει προσαρμογή με τι εξελίξει και του αναγκαίου ρόλου του νομοθέτη να προβάλλει αντιρρήσει και να απορρίπτει ή να εγκρίνει τι προτάσει. Λοιπόν, ε, ε, καλωσορίζω σχόλια, προτάσεις, συνάδελφοι, ειδικά σας σχόλια και προτάσεις όσον αφορά το σχέδιο προκατατικής εκθέσεως που υπέβαλα και προφανώς όπως προανέφερα είμαι ανοιχτή προς συζήτηση και βεβαίως θα διοργανωθεί και μια συνάντηση με τους Κιώδης τώρα που έχουμε επιτραπέζης έκθεση για να δω τι τροπολογίες θα θέλετε να υποβάλλετε. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ Αρλίν. Είχαν πρόβλημα οι διερμηνείς και έβλεπα πολλά κόκκινα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Δεν είναι εδώ ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. Βίκη, θες να πάρεις εσύ το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική νομοθεσία. Όχι μόνο για αυτά που κάνει αυτά καθ' αυτά, αλλά και γιατί στέλνει ένα μήνυμα για το ποια είναι η άποψη του Κοινοβουλίου για αυτά τα θέματα. Αλλού μιλάμε για νομοθετικές πράξεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον ή για το πώς θα μπορούσαν να είναι οι ελεκτικές αρχές στο μέλλον. Εδώ όμως μιλάμε για δράσεις που ζητάμε να ληφθούν τώρα, αμέσως. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό θέμα όλη η γλώσσα που έχουμε χρησιμοποιήσει καλύτερο ρυθμιστικό περιβάλλον, καλύτερη διακυβέρνηση κτλ. Όλα αυτά εφαρμόζονται με αυτήν την πρόταση. Αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για τις τράπεζες όταν μιλάμε... Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε και προηγούμενες ε, διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει για να καταλάβουμε από πού προέρχεται αυτή η διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει γίνει καλός καλή ανάλυση αντικτύπου. Έγινε πέρυσι εν μέρη στη Βασιλεία για τμήμα της ε, εμπορικής κεφαλαιοποίησης γιατί ζητάμε αύξηση της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέχρι το 2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Μετά όμως στη Βασιλεία άρχισαν να εξετάζουν ένα θέμα συσχέτιση συναλλαγών και μετά ζητήθηκε νέα ανάλυση αντικτύπου με εκατοντάδες ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν και κατέληξαν σε μία έκθεση τον Ιούνιο. Άρα, οι επιπτώσεις μπορούν να είναι πολύ σημαντικές. Και πολύ σημαντικά είναι και τα νούμερα που μας δίνουν οι τράπεζες, όπως επίσης και τα νούμερα που μας δίνουν κάποιες ρυθμιστικές αρχές. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Σιγκαπούρη ανησυχούσαν πολύ για το θέμα η Fed και άλλες τράπεζες. Όμως υπάρχει συνένεση ότι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη κεφαλαίο, κεφάλαιο οι τράπεζες για τις πράξεις ε, επανατυκλοποίησης και για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Και να σας πω τι είπε ο Λόρδος Μάντελσον, πρώην επίτροπος. Πριν από δύο εβδομάδες μιλούσε σε μεγάλες επιχειρήσεις και είπε για το κεφάλαιο πρέπει να εφαρμοστούν νέοι κανόνες με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο χρονοδιάγραμμα που να μην δημιουργεί αβεβαιότητα σήμερα και που να μην δυσκολεύει τις τράπεζες στο να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Συμφωνώ απολύτω μαζί του. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Κάποιες τράπεζες λένε ότι αυτή η νομοθεσία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δυνατότητά τους να δίνουν δάνεια. Και ακούσαμε και τον κύριο Στοσκάν το πρωί που να λέει ότι πρέπει να αυξήσουμε την ιδιωτική χρηματοδότηση τώρα. Γιατί έχουμε και το όραμα για το 2020 με την ε, απανταχού ευρυζωνική σύνδεση την ενεργειακή ασφάλεια κτλ. κτλ. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα χρειαστούν τραπεζική χρηματοδότηση. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε και την πλευρά των τραπεζών και δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει καλή ανάλυση αντικτύπου. Και δεν νομίζω ότι η Επιτροπή μας έκανε καλός που δεν έκανε καμία ακρόαση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ακούσω και τις ανησυχίες της ΦΕΔ, η οποία δεν εφάρμοσε ποτέ τη Βασιλεία 2. Θέλω να έρθουν εδώ και να τους πούμε εμείς, εμείς προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Θα συμπορευτείτε. Επίσης θα ήθελα να ακούσω κάποιες από τις μεγάλες τράπεζες, αν έχουν παραπονεθεί, να παραπονεθούν δημοσίες για τις συνέπειες από τις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αν λοιπόν πρόκειται να αυξήσουμε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις πρέπει να έχουμε αποδείξεις για το αν μπορούν ή όχι να ανταποκριθούν σε αυτή την απέτηση τώρα. Γι' αυτό θα έπρεπε να ζητήσουμε να ακούσουμε την άποψή τους. Η συγγήτρια μας είπε ότι πρόκειται να ακούσει ανεξάρτητες ε, περιπτώσεις με καλά επιχειρήματα. Θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό και ενδεχομένω θα έπρεπε να ακούσουμε και κάποιους μη ανεξάρτητους. Αλλά να ακούσουμε τα επιχειρήματά τους. Πριν η Αρλίν μίλησε για χειροπέδες και για αλεξίπτωτα. Είναι διαφορετικά αυτά τα δύο. Τώρα, άμα θέλουμε να δούμε την γενικότερη εικόνα. Γιατί μιλάμε μόνο για Ευρώπη, αφού το θέμα αφορά και πέρα από τους G20. Γιατί μόνο οι τράπεζες. Δεν ξέρω, αυτά αναφέρονται και στις τροπολογίες μάλλον. αν τα κράτη-μέλη θέλουν να πάνε πέρα από το G20, για τις αμοιβέ, αυτό θα έπρεπε να είναι εθνική απόφαση, όχι ευρωπαϊκή απόφαση. Γιατί τέτοιου είδους αποφάσεις επηρεάζουν και τις δυνατότητες φορολόγησης των κρατών μελών και άρα θα έπρεπε να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να πούν την άποψή τους. Ευχαριστώ, Πασκάλ. Η ερμηνεία μας είναι μάλλον ε, θετική όσον αφορά το πακέτο που προτείνει η Αλήν Μακάρθη. Καταρχάς ε, όσον αφορά τις αμοιβέ, ε, το γεγονός ότι δίνεται δυνατότητα κειμενόμενων αμοιβών για όσες, για όσες τράπεζες έλαβαν ε, βοήθεια, ενίσχυση, καθώς και το γεγονός ότι θα υπάρχουν κάποια όρια Νομίζω ότι είδαμε ότι μετά από αυτά που υπόθηκαν από το G20 πριν από ένα χρόνο, δημιουργήθηκαν κάποια περισσότερα εργαλεία από τις τράπεζες για τον έλεγχο της κατάστασης και αυτό θα έπρεπε να αναφερθεί. Όσον αφορά τις ε, κειμενόμενες αμοιβές, ε, τα bonus, θα ήθελα να ρωτήσω αν ε, αναφέρεται εκεί και το πακέτο αμοιβή ε, όταν κάποιος ε, παρετείται ή διακόπτει τη συνεργασία. Θα έπρεπε να είναι πιο σαφής ο ορισμός του μπόνους προκειμένου να γνωρίζουμε ακριβώς που αναφέρεται. Τώρα κάποια άλλα θέματα που αναφέρονται στις τροπολογίες. Καταρχάς όσον αφορά την ε, περίπλοκη τιτλοποίηση και τις πράξεις επανατιτλοποίησης. Κανείς δεν γνωρίζει τι είναι αυτά, και κανείς δεν μπορεί να αξιολογήσει πλήρως τους κινδύνους. Άρα έχουμε δύο δυνατότητες. Εμπιστευόμαστε τις τράπεζες για να κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις και να ενημερώσουν τις ρυθμιστικές αρχές ή λέμε ότι αυτό το παιχνίδι το παίξαμε στο παρελθόν και είδαμε που καταλήξαμε. Μας ενδιαφέρει να μειώσουμε τους κινδύνους και να δημιουργήσουμε αρκετούς περιορισμούς προκειμένου οι τράπεζες να μην μπαίνουν στον πειρασμό να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα των οποίων δεν έχει αποδειχθεί το όφελος για την οικονομία, την πραγματική οικονομία για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης διαπιστώνω ότι από τότε που ξεκίνησαν αυτά τα προϊόντα, τέλη της ε, δεκαετίας του 90 περίπου, μειώθηκε και η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ενώ παλαιότερα που είχαμε ένα απλούστερο και λιγότερο περίπλοκο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί οι τράπεζες να πήγαιναν χειρότερα στην Ευρώπη αλλά είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη δηλαδή με, ένα, με απλούστερα προϊόντα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια μειώθηκε η ανάπτυξη και διαπιστώσαμε και ποια ήταν τα προβλήματα, ποιοι ήταν οι κίνδυνοι για το σύνολο της οικονομίας από αυτές τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οπότε, ακόμη και αν δεν το κάνουν άλλων, νομίζω ότι θα ήταν εποφελές να έχουμε ένα πιο απλούστερο, ένα πιο απλό και πιο εύκολα αξιολογήσιμο σύστημα. Και δεν νομίζω ότι θα χάσουμε πολλά αν ελέγχουμε περισσότερο τις διάφορες ε, πράξεις πολύπλοκης τυκλοποίησης που θα έχουν στη διάθεσή τους οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Να πω κάτι άλλο τώρα. Αυτή τη στιγμή τέσσερις τράπεζες μόνο από όλες τις ευρωπαϊκές ασκούν δραστηριότητες ε, τις οποίες προσπαθούν μέσω Λόμπιν να διατηρήσουν. Εμείς όμως θα έπρεπε να αποστασιοποιηθούμε από αυτό το Λόμπιν και να εξετάσουμε και αυτού του είδους τα εργαλεία και να διαπιστώσουμε αν όντως ε, έχουν περισσότερα θετικά από ότι αρνητικά στοιχεία και να μην διστάσουμε αν διαπιστώσουμε το αντίθετο να εφαρμόσουμε πιο αυστηρούς κανόνες τουλάχιστον μέχρι να έχουμε νέες αναλύσεις αντικτύπου γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα μικρό μερίδιο της αγοράς που αφορά μόνο τέσσερις τράπεζες που κάνουν αυτές τις ιδιαίτερα περιπλοκές Ευχαριστώ εγώ με σκιώδη συγγήτρια για την Άλτε, οπότε θα προσπαθήσω και εγώ να μιλήσω και να ακολουθήσω την ίδια σειρά όπως η συγγήτρια. Λοιπόν, καταρχάς ερχόμαστε στο ενδιαφέρον θέμα των αμοιβών και των πόνους και σήμερα το πρωί ακούσαμε τον Μάριο Ντράγκη που αναφέρθηκε γενικόλογα στα ευκταία μετά την χρηματοσυντική κρίση. Είπε ότι πέρα από το συμπληρωματικό ε, κεφάλαιο δεν θέλαμε αρνητικά κίνητρα να δοθούν. Αυτός ήταν ο στόχος μας σε αυτό το κομμάτι του κειμένου. Κανείς δεν φαίνεται να υπογράμμισε ότι μπορεί ίσως να είναι αρνητικό κίνητρο οι μετοχές, διότι είναι ένα κίνητρο για κέρδη ε, εγγενές. Δηλαδή θέλει κανείς να πάρει μερίσματα. Άρα τι κοιτάμε εδώ, τι βλέπουμε. Αν πούμε ότι θέλουμε να φροντίσουμε για την κοινωνία εν γέννη, πέρα από τα κέρδη, τότε δεν επιλύεται το πρόβλημα αν τα μπόνους καταβάλλονται κυρίως σε μετοχές παρόλο που θα προβλέπετε περίοδους που δεν μπορούν να α, πρέπει να κρατηθούν. Είναι μερική κάλυψη του θέματος αυτή. Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Και μου αρέσει η ιδέα που αναφέρεται. Δηλαδή χρήματα του μπόνους να μπαίνουν σε ένα κεντρικό κουμπαρά αν θέλετε και μένει εκεί και μετά αργότερα μπορεί να πάρει κανείς τον πόνους αν όλα πάνε καλά. Και θα πρέπει να δούμε και το θέμα της συνολικής αμοιβή. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι κάτι είναι ένα ποσοστό του βασικού μισθού, διότι ξέρουμε τι συμβαίνει με τον βασικό μισθό. Αυτό που συνέβη στι Ηνωμένε Πολιτείε, όταν προσπάθησαν να μειώσουν, να περιορίσουν τα μπόνους και πριν. Άρα θα πρέπει να πούμε κάτι για τη συνολική αμοιβή. Δεν είμαι σίγουρη ε, για το πώς θα, θα καλύψουμε και τα συνταξιωτικά ποσά, μία. Εγώ θα ήθελα να εξετάσουμε το θέμα περαιτέρω. Μ' άρεσε η ιδέα της βαθμονόμησης διότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε με ένα άλμα να προχωρήσουμε ως εκεί που θα ήθελα, ίσως μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μέσω της ιδέας της βαθμονόμησης. Θα ήθελα να το εξετάσουμε περαιτέρω, να το συζητήσουμε με τους κοιόδης και με άλλους. Ανακοινώθηκε ένα πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο μπόνους από πλευράς ε, Deutsche Bank, ε, άρα δεν βοηθούν τον εαυτό τους οι τράπεζες. Κάποια ανώτατα στελέχη ε, συγκρατήθηκαν βέβαια στο κάτω μέλος που γνωρίζω καλύτερα. Και εγώ ανησυχώ όσον αφορά το γενικό αντίκτυπο όλων αυτών. Δεν μιλάμε μόνο για τον αντίκτυπο αυτής της οδηγίας. Έχουμε πολλά άλλα θέματα και αλλάζει και ποιο είναι, τι θεωρείται το βασικό κεφάλαιο. Το υβρίδιο κλπ δεν είναι διαθέσιμα. Μεγάλες αλλαγές ήδη έχουν δρομολογηθεί και από το CRD2. Εγώ δεν διατείνομαι ότι συστήνω μεγάλη καθυστέρηση, αλλά ήδη έχει προγραμματιστεί εργαστήριο ή μια ακρόαση σχετικά με το πρόγραμμα υπαριθμών 4 και τη ρευστότητα. Και διαρωτώ με, μήπως μπορούμε να κάνουμε πιο εκτεταμένη ακρόαση Πρέπει να το συζητήσουμε αργότερα με τους συντονιστές αυτό. Θα πρέπει να προσέξουμε κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε το σωστό συνδυασμό. Ίσως να είναι δύσκολο οργανωτικά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ψηφοφορίες, τις ακουράσεις κλπ. Εγώ είμαι πρόθυμη όμως να προσπαθήσω. Αν χρειαστεί, γιατί να μην αλλάξουμε λίγο το χρονοδιάγραμμα μας, να το μετακινήσουμε κατά ένα μήνα για να, κάνουμε, να καλύψουμε τις ευρύτερες αξιολογήσεις ε, συνεπιών της Βασιλείας και του FSB. Θα ήταν καλό να τα έχουμε αυτά πριν από την ψηφοφορία στην Επιτροπή, αντί του να καταφθάνουν αυτά τα πορίσματα εν μέσω τριμερούς διαλόγου. Αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια προσαρμογή, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε δημοσία γιατί το κάναμε. Υπέχουμε υποχρέωση να είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται. Αυτές οι κρίσιμες αποφάσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνονται εντός τριμερούς διαλόγου. Βέβαια θα αποκαλυφθεί η τελική απόφαση, αλλά όχι τα επιχειρήματα που ανταλλάχθηκαν και ποιος είπε τι. Για ένα μήνα τώρα, περίπου, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πιεστούμε και να κάνουμε λάθος. Ίσως να μπορούμε να βάλουμε στις ανατεθήσεις πράξεις κάτι. Είχαμε και ένα εργαστήριο όσον αφορά τη φερεγγιότητα 2 για τα εφαρμοστικά μέτρα αυτού. Χθες συμμετείχαν όπως και υποφαινόμενοι σε αυτό. Και εκεί επί μακρόν υπήρξε το εξής πρόβλημα. Παλεύαμε με τα εφαρμοστικά μέτρα που προτινόταν. Θεωρούσαμε ότι ίσως ξεπερνούσαν αυτά που καθορίσαμε για το επίπεδο 1 και έπρεπε να διώξουμε αρκετά από αυτά τα μέτρα. Τουλάχιστον τώρα πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν διαβάσετε τις εφημερίδες, θα δείτε ότι έγιναν προτάσει επιτροπή επίπεδου 3 που εθετούσαν στάσεις ή προτάσεις που ήταν τοποθέτηση διαπραγματευτική. Και εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν σε αυτές τις επιτροπές που με την πάροδο του χρόνου θα γίνουν υπηρεσίες με τεράστιες εξουσίες. Και δεν θέλω να ασκούν τέτοιου είδους εξουσίες επί διαπραγματευτικής βάσεως. Δεν το θεωρώ σωστό. Αυτές τις ανατεθήσεις πράξεις, εχωρηθήσεις πράξεις πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε πάντα τη δυνατότητα να αρνηθούμε. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο με το πηγενέλα στις συζητήσεις για την βασική πράξη. Εάν εκχωρούμε πολλά στις εκχωρηθήσεις πράξεις δεν είναι και πολύ σωστό. Όσον αφορά το, το θέμα της επανατιτλοποίησης που είναι πολύ περίπλοκο δεν κατάλαβα γιατί το κάναμε ήδη στο CRD2 είχαμε απαιτήσει για τη σωστή προσέγγιση και προσοχή και αν δεν συμμορφώνονται με αυτό πάμε στο τέλος το κεφαλοχικό ένα προς ένα και είναι θέμα αναλογικότητας. Αν υπάρξει ε, κάποιο μικρό προβληματάκι υπάρχει αναλογική προσέγγιση. Αναλογικότητα όμως σημαίνει εξέταση και της περιπλοκότητας ενός ζητήματος. Αυτό που λέει από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι μέχρι ότου αποδειχθεί στην αρμόδια αρχή ότι έχουν συμμορφωθεί με τις ίδιες απαιτήσει για τη σωστή προσέγγιση που ήδη προβλέπεται σύμφωνα με το CRD2, ότι έχουν αυτό το κεφαλουχικό τέλος ένα προς ένα. Άρα δεν βλέπω τι νόημα έχει αυτό. Κυρίως όταν κανείς δεν μπορεί να καθορίσει τι εννοείται εδώ με την αποτιτλοποίηση, επανατιτλοποίηση μάλλον. Είναι εντός του χαρτοφυλακίου που οριμάζει και αντικαθίσταται. Διότι αυτό συμβαίνει. Μερικά από, όλα αυτά, μερικά από αυτά είναι δυναμικής φύσεως και επειδή είναι δυναμικά ίσως είναι πιο αναγκαίο να εντοπίζουμε το, το δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό έχουμε αυτέ τι απαιτήσει στην προσέγγιση του CRD2 για να αντιμετωπίσουμε αυτό το δυναμικό χαρακτήρα. Το Συμβούλιο νομίζω ότι καλά το έκανε και διέγραψε αυτή την απέτηση. Και εγώ τι άλλο θα ήθελα να κάνω. Να βάλουμε ρήτρα αναθεώρηση. Όπω κάναμε και για την τυπλοποίηση στο CRD2. Είπαμε, α δούμε πώ πάνε τα πράγματα και ας κάνουμε κάτι υπό το φως της εμπειρίας. δεν είναι πλεονασμός μόνο. Απαιτείται ορισμός κάποιου στοιχείου που ίσως τελικά οδηγήσει σε απροσδόκητες συνέπειες. Κάτι επιζήμιο. Αν κάναμε ακρόαση, θα εξετάσαμε και για το εμπόριο συσχετισμού. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για αυτά και ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος του να καθορίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο. Ξέρω ότι δεν θέλατε να καθορίσουμε ένα κατώτατο όριο, αλλά θα ήταν καλό να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε και πέρα του να λέμε ότι μπορεί να γίνει αυτό με εκχωρηθήσα πράξη, ανατεθήσα πράξη, ίσως θα μπορούσαμε να θέσουμε και άλλους περιορισμούς εντός αυτής της ανάθεσης. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που έχω να θίξω. Η Σιλβή Γκουλάρ είναι η επόμενη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μακάρτη, για τη δουλειά που έκανε. Είναι αρκετά γενναία που ενεβάθυνε σε ένα θέμα που παρέμεινε ε, μη αναλυμένο επί οι φυσικέ ρήτε διαφύλαξη εντό των επιχειρήσεων, των εθνικών συστημάτων και λεφτά επιφεύγουν να αποφευτούν οι καταχρησοφάτα μπόνου, αλλά η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δείχνει ότι υπήρξαν καταχρήσει και θέλω να πω στη Βίκη ότι είναι αρκετά ενοχλητικό. Θα έπρεπε να γίνουν μελέτες αντικτύπου για να προστατευτούν εκείνοι που ζουν καλά και στην ανάληψη του κινδύνου όταν υπάρξει σε, που έχουν μεγάλη συνέπεια αυτέ οι ανήψει κινδύνου χωρί να τι μελετούν. Το βάρο απόδειξη θα ήταν καλό να μην είναι πάντα προ την πλευρά εκείνων που δεν έκαναν τη ζημιά. Τρει παρατηρήσει έχω. Η πρώτη, όσον αφορά αυτό το θέμα που θα συμπεριλαμβάνεται σε όλε τι εκθέσει και το είδαμε όλο το πρωί. Περιμένουμε του Αμερικανού ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Κάνουμε πράγματα μόνοι μα ή όχι. Και εκεί πιστεύω ότι μπορούμε δύσκολα να υποστηρίξουμε ταυτόχρονα ότι η καλή λύση είναι παγκόσμια, γενική και η λήψη γενική λύσεω θα κινηθούμε σε εθνικό επίπεδο. Από την πλευρά μου, όπω είπε και η συγγήτρια, θεωρώ ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα άλλα τα κάλυψαν άλλοι συνάδελφοι, αλλά η ιδέα περιορισμού της βαθμιαίας αμοιβή του είναι κάτι πολύ λογικό για να αποφευθεί ο κίνδυνος αφήνοντα δυνατότητε επιχειρήσεις επιχειρήσει να αποφασίσουν αύξηση τη αμοιβή ε, τη βασικού μισθού των, μας, των μισθωτών και κατά πόσο σχετίζεται με την ανάληψη κινδύνων. Τελευταίο σχόλιο. Δεν τρομάζω από την ιδέα σύμφωνα με την οποία οι αρχές, που, η αρχή που δημιουργούμε, οι αρχές που δημιουργούμε λέγω, να δημιουργηθούν βάσει βαθμολόγησης, βαθμονόμησης. Είναι καλή ιδέα ή να συμμορφώνονται με άλλα σημεία. Αν θέλουμε να υπάρχει εποπτεία, θα πρέπει αυτέ οι αρχέ να μπορούν να δουν και να ελέγχουν και να βαθμολογούν τι συμβαίνει στι επιχειρήσει. Αυτά και ευχαριστώ. Okay, I, I think that that uh, Vicky wanted to reply to some of those things about. Η Vicky θέλει να απαντήσει για κάποια πράγματα για την ε, μελέτη επιπτώσεων, αυτό ίσως στο τέλος. Ο κύριος Κλούτ. Ο Γιώργεν παρακαλώ. yes. Νομίζω ζήτησε να παρέμβει. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα μια σκέψη, μια πρόταση από πλευρά Πασκάλ να αναφέρω. Πολύ σωστά κιόλα ανέφερε πιστεύω ότι η απορρίθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών τα τελευταία δέκα χρόνια δεν συνεισέφερε στην ανάπτυξη, όμως κέρδισαν πάρα πολλοί τράπεζες ε, σε σχέση με μια ανακατανομή όσον αφορά την κοινωνία, πράγμα που θα πρέπει να το δούμε με κριτικό πνεύμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Από αυτό εξαρτάται και η αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους πολίτες μας. Πολύ καλό αυτό σε σχέση με αυτή την γενική, κατάσταση πραγμάτων. Μία παρατήρηση όσον αφορά τις αμοιβέ ε, και τα πριμ. Γενικά, απλά συμβαίνει το εξής. Πολλοί πολίτες, σαν συνέπεια αυτής της κρίσης, βλέπουν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται. Σαν συνέπεια της ανεργίας χάνουν εισόδημα, περικόπτονται τα εισόδηματά τους. Έχουμε και τη συζήτηση όσον αφορά το πρόβλημα της Ελλάδας. Αυτοί οι πολίτες στην Ευρώπη βλέπουν ότι με περιορισμό των χρημάτων τους, των εισοδημάτων τους πληρώνουν τα σφάλματα των τραπεζών και του οικονομικού συστήματος. Εκείνοι πληρώνουν τα σπασμένα ως αντιστάθμιση και θα δουν πάρα πολύ κοντά τι κάνουμε σε σχέση με τις αμοιβέ και τα πρίμια της τράπεζες. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να βρούμε μια ευφυή, μια καλή λύση για τον περιορισμό αυτών των ε, εισοδημάτων και το λέω συνειδητά πρέπει να υπάρξει περιορισμός των απολαβών αυτών των ατόμων. Αυτό συνεισφέρει σημαντικά οι πολίτες να θεωρούν αποδεκτό το σύστημα, κοινωνικά αποδεκτό όταν είναι δικαιότερο με περικοπή τέτοιων αμοιβών. Αυτό από πλευράς ε, αποδοχής είναι σημαντικό στοιχείο, να το δούμε πώς επιδρά στους πολίτες. Θα εξαρτηθεί από εμά να βρούμε ικανοποιητικέ λύσεις, να λύσουμε το πρόβλημα αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά, από πολλούς πολίτες θεωρείται σκανδαλώδη η κατάσταση. Ότι εκείνοι που συνεισέφεραν σημαντικά στην δημιουργία αυτής της χρηματοοικονομική κρίσης, αυτή τη στιγμή πάλι σχετικά <clears throat> αυρόχης ποσοί πέρασαν το ποτάμι. Και μάλιστα όχι μόνο χωρίς πρόβλημα, αλλά κέρδισαν και έτσι δεν συμμετέχουν στη χρηματοδότηση της κρίσης, των ζημιών της κρίσης με κανέναν τρόπο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα ρυθμίσουμε και ως γκουε θα υποβάλουμε τροπολογίες και εμείς. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει από πλευράς πρότασης και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Θα έχουμε τροπολογίες που θα καταθέσουμε εμείς. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και να καθυστερήσουμε. Ένα πράγμα θέλω να πω, επειδή το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο και αυτό και οι παρεμβάσει των προλαλισάντων και προλαλισσασών το έδειξαν. Νομίζω ο τρόπος με τον οποίο για την μεθοδολογία κάνω τώρα λόγο, έτσι, για την μέθοδο προσέγγισης και εργασίας, μεθοδολογία της εισηγήτριας θέλω να αναφερθώ. Ο τρόπος με τον οποίο προχωρεί η Αρλίν εδώ, δηλαδή σε ένα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα <clears throat> να πει ότι θα κατευθυνθώ προς αυτή την πορεία, σε αυτή την κατεύθυνση με συνέπεια γιατί θέλω να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και με συνέπεια αλλά θα είμαι ανοιχτή για στοιχεία που θα υποβληθούν σε μένα για ανεξάρτητες ε, ρυθμίσεις. Δηλαδή δεν είναι ας το πω έτσι πληροφορίες ε, από τις επιχειρήσεις ε, ε, προκατηλημένες αλλά αντικειμενικά επιχειρήματα και υπό αυτού του είδους αντικειμενικά επιχειρήματα είμαι πρόθυμη να κάνω τροπολογίες και να αλλάξω την πρότασή μου. Εξαιρετικό αυτό διότι ακριβώς εκεί όπου πάρα πολύ τεχνικά θέματα αντιμετωπίζουμε η σωστή πορεία είναι αυτή. Δηλαδή για την Επιτροπή μας <clears throat> να εργαστούμε για τη μεταρρύθμιση με σαφή πορεία και ανοιχτό πνεύμα. Υποστηρίζω λοιπόν σε σχέση με τους συναδέλφους που έχουν κάποιες άλλες απόψεις σε λεπτομέρειες <clears throat> με αυτή τη μέθοδο να μπορέσουμε να εργαστούμε και έτσι να προσαρμοστούμε. Γιατί έτσι μπορούμε ένα λογικό ευφυές προϊόν ε, σκόπιμα να παράξουμε. Εδώ πρόκειται και για θέματα ακροάσεων που όπως εσείς πρόεδρε λέτε ότι έχει νόημα <clears throat> να έχουμε πρόσθετη πραγματογνωμοσύνη που θα χρειαστούμε αν αυτό δεν οδηγήσει σε μεγάλη καθυστέρηση των εργασιών μας, λογικό και σκόπιμο είναι αυτό. Κανένας δεν είναι εναντίον πρόσθετης πραγματογνωμοσύνης ε, ως στοιχείο υποστήριξης που μπορούμε να έχουμε. Και επιπλέον θέλω να πω, παρότι προσπαθώ να έχω τη δική σας άποψη και να ευθυγραμμίζομαι, στο θέμα αυτών των περίπλοκων θεμάτων μπορεί κανείς να έχει και μια διαφορετική άποψη βλέπει κανείς την ανάγκη να ρυθμιστούν τα πράγματα, αλλά μπορεί να επιλέξει μια άλλη κατεύθυνση προς τη ρύθμιση. Αλλά αυτό οι διαβουλεύσεις μας θα το δείξουν πώς πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Βίκη ε, έκανε ό,τι μπορούσε για να σηκώσει η γαλάζια κάρτα ή ό,τι πιο κοντινό βρήκε. Να σας δώσω το λόγο λοιπόν. Κοιτάξτε, έχουμε υπέροχους μεταφραστές, αλλά άκουσα τη Σιλβή να αναφέρει το όνομά μου. Αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς τι είπε. Όταν αναφέρεται κάτι προσωπικό θα ήθελα να καταλαβαίνω ακριβώς τι έχω, υποτίθεται έχω πει. Άκουσα το όνομά μου κάποια αναφορά και δεν άκουσα τι υποτίθεται τι είπα. It was about the impact assessments and thank you very much for suggesting that you could maybe tidy that up into CRD4. Λοιπόν, θέλαμε αυτά να εντάξουμε στο CRD4 όσον αφορά τη μεικτή ακρόαση. Και δεν υπήρξε συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών για λόγους χρονικούς. Θα ήταν καλό να γίνουν κάποιες συναντήσεις πριν την προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Θα βοηθούσε πολύ, όπως έχουμε ξανακάνει. Και εφόσον έχω το λόγο να πω κάτι άλλο για την πολύ το περίπλοκο θέμα, πολύ περίπλοκο θέμα ...το της τυπλοποίησης. Πώς καθορίζουμε τι είναι πολύ περίπλοκο. Κάτι που είναι κάτι πολύ περίπλοκο για ένα θεσμικό όργανο, ίσως να μην είναι για κάποιο άλλο. Όπως και σε άλλους τομείς της αγοράς, ας πούμε επαγγελματικοί, οι επαγγελματίες επενδυτές αντιμετωπίζουν διαφορετικά από ότι οι μη επαγγελματίες επενδυτές. Κάποιοι επενδυτές δεν έχουν το επίπεδο τη γνώσης να αντιμετωπίσουν κάτι που είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλοι Απ' την άλλη πλευρά θα περίμενε κανεί οι Λίμανς να καταλάβαιναν κάποια πιο περίπλοκα θέματα περί τυπλοποίησεων από ό,τι έκαναν. Είτε μπορεί να πει CRD2 να δούμε αν λειτουργήσε, είτε, είτε να προσπαθήσεις να διαφοροποιήσει την περιπλοκότητα και τη διαφοροποίηση μεταξύ επαγγελματιών μη επαγγελματιών. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι υπάρχουν διάφορε προσεγγίσεις. Δεν άκουσα το όνομά σου, Βίκη. Δεν είμαι σίγουρη, λέει η πρόεδρο. Τέλο πάντων. Να δώσω το λόγο στη Σιλβή. Αλλά ένα σχόλιο που είχα στον αφορά τι αξιολογήσει αντιχτύπων ήταν ότι δεν ζητάμε μόνο αξιολογήσει αντιχτύπων για τι τράπεζε. Δεν είναι αυτό που υποστηρίζουμε, αλλά πιο πέρα. Θέλουμε να δούμε ποιε είναι οι συνέπειε στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι κάτι που έχουμε στην καρδιά μα. Αυτό είναι το κλειδί που θέλουμε να εξετάζουν οι ε, αξιολογήσει συνεπιών. Το είπε και ο Μάριο Ντράγκη το πρωί. Σιλβί, ακριβώ ήθελα να πω κάτι τυπικό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πολύ περιεκτική και συνοπτική η Γαλλία. Δεν αναφέρθηκα εγώ στο ΣΥΝΤΕΑ 3 και στο 4. Εγώ είπα μόνο ότι εξεπλάγει από του ελιγμού που μπορεί να καθιστέσουν τα πράγματα βάσει τη ιδέα ότι θα πρέπει πάντα να μελετούμε τι συνέπειε όσον αφορά την πραγματική οικονομία των κειμένων μα. Ενώ Εκείνοι που πλήττονται από αυτούς τους νόμους δεν εξετάζουν ε, πώς η συμπεριφορά τους η πολύ παρακινδυνευμένη επηρεάζει και πλήττει την πραγματική οικονομία. Αυτό ήταν που ήθελα να πω και ευχαριστώ. I think Γι' αυτό προσπαθούμε να τους τιμωρήσουμε λίγο. Νομίζω ότι μίλησαν όλοι όσοι ήθελαν το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ετέθησαν πολλά θέματα, κάποια θα τα συζητήσουμε διμερώς ή στην άντιση των σκιωδών εισηγητών. Τώρα, για τα σχόλια που έκανε η Βίκη. Πολλοί ζήτησαν αναλύσεις αντικτύπου. Ορισμένοι γιατί όντως θέλουν να διαπιστώσουν αν όντως πρόκειται να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Ορισμένοι ζητούν ανάλυση αντικτύπου απλά για να ευδραδίνουν τη διαδικασία. Και τα περισσότερα από τα επιχειρήματα που ανέφερες τα άκουσα από τα λόμπι των τραπεζών. Γνωρίζω ότι όντω πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και με τις ανησυχίες των τραπεζών αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να υπάρξει κάποια ισορροπία. Και δεν είναι σωστό ότι δεν έχουν γίνει αναλύσεις αντικτύπου. Έχουν γίνει και έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε νέες αναλύσεις αντικτύπου επειδή αυτό θέλουμε να κάνουμε. Εγώ επαναλαμβάνω, είμαι ανοιχτή. Αν όντω υπάρχουν πραγματικά προβλήματα για την πραγματική οικονομία, όντω θα τα εξετάσουμε. Όμως αυτή τη στιγμή οι ανησυχίες των τραπεζών δεν αφορούν τόσο το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τις επανατιτλοποιήσεις, αλλά το CRD4 γιατί θεωρούν ότι το CRD4 δημιουργεί περισσότερες λεπτομέρειες από ότι το CRD3 και θέλουν να το δουν με περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, αυτό που είπες για τον Λόρδο Μάντελσον ήταν λίγο προβληματικό. Συζητάω συχνά με τον Λόρδο Μάντελσον και ε, μέσω τηλεφώνου και από κοντά και ήταν σαφής ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομείου και ότι χρειαζόμαστε για σταθερό τραπεζικό σύστημα και μάλιστα στην ομιλία του μιλούσε για τον σορευτικό αντίκτυπο μια σειρά μέτρων, όχι μόνο για τα sdr3. Κανείς λοιπόν, ούτε και η Ισπανική Προεδρία δεν ζητάει καθυστέρηση της εφαρμογής αυτών των προτάσεων. Παρόλο που βεβαίως επαναλαμβάνω θα εξετάσουμε θέματα που όντως χρήζουν εξέτασης. Τώρα όσον αφορά τις αμοιβέ, είπε η Βίκη Φόρντ ότι πάμε πολύ μακριά. Κοιτάξτε τις ε, προτάσεις μας. Δεν πηγαίνουν μακρύτερα από τις προτάσεις του G20. Βεβαίως είναι και θέμα διερμηνίας, με συγχωρείτε αυτό. Όμως, γιατί προκύπτει το πρόβλημα με τις τράπεζες. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι οι τράπεζες ε, σχεδόν κατέλεξαν σε κατάρρευση του κόσμου εξαιτίας των πόνους και των αμοιβών τους. Αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος της ύφεσης, αυτό πιστεύει το κοινό, ακόμη κι αν εσύ διαφωνείς. Οπότε... Πολλοί αναρωτιούνται για το αν γίνει κάτι στην Ευρώπη, αν θα γίνει αυτό και στην Αμερική σε άλλες χώρες. Αυτό που βλέπουμε από τις προτάσεις του G20 είναι ότι αρκετές χώρες θα κάνουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, ενδεχομένως όχι την ίδια στιγμή. Αλλά αν δείτε τι προτείνεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική, υπάρχουν προτάσεις που είναι ακόμη πιο αυστηρές από αυτές που προτείνουμε στην Ευρώπη και υποθέτω ότι και κάποιοι από τους συναδέλφους θα κάνουν προτάσεις ακόμη πιο αυστηρές και προς την ίδια κατεύθυνση που κινούνται οι αυστηρές προτάσεις στην Αμερική. Πολύ γρήγορα, λέει η Πρόεδρος. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τις αμοιβέ και τα μπόνους. Ο λόγος που κάνω αυτή την πρόταση και επαναλαμβάνω ότι δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η ιδανική λύση η τελευταία μου λήξη αλλά λέει και η FSRB ότι πρέπει να έχουμε ισορροπία και αναλογικότητα. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε ισορροπία και αναλογικότητα αν το 90% της αμοιβή είναι τα μπόνους. Όσον αφορά τις μετοχές, Συμφωνώ ότι ναι, ακόμη και όταν λαμβάνετε τα μπόνους σε μετοχές, πάλι έχετε κίνητρα για ανεπίτευξη κίνδυνους, όμως παράλληλα έχετε συμφέρον για τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη απόδοση της τράπεζας. Γιατί το πόνου σας θα εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη απόδοση της τράπεζας. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και άλλες προτάσεις. Για παράδειγμα, πόνους με τη μορφή συντάξεων Όσον αφορά τώρα τις επανακυκλοποιήσεις, είναι κάτι που πρέπει να επανεξετάσουμε. Όπως είπε η Σάρων, ήδη μας απασχολεί το θέμα στα πλαίσια του CRD2. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλήξει σε τελική άποψη, αλλά αποφάσισα και ευχαριστώ τον συντονιστή που με κατανοεί Αποφάσισα λοιπόν ότι εφόσον δεν έχουμε αποδείξεις δεν πρόκειται να προτείνω αλλαγές. Εκτός αν μου δείξετε αποδείξεις ή αναλύσεις αντικτύπου που να οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτά από εμένα και να υπενθυμίσω κυρία Πρόεδρε ότι είχαμε ζητήσει ακρόαση για αυτή την πρόταση. Όμως επειδή έχουμε πολλά θέματα που χρήζουν ακροάσεων είναι δύσκολο να τις διοργανώσουμε όλες. Οπότε είναι ένα ερώτημα το αν πρέπει να έχουμε δύο ακροάσεις για τα CRD, όσο σημαντικά και να είναι αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να κάνουμε ακρόαση για ορισμένες μικρές τεχνικές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Νέες ημερομηνίες αν και μπορεί και πάλι να αλλάξουν λίγο. 25 Μαρτίου κατάθεση τροπολογιών, εξέταση τροπολογιών 26 Απριλίου, με στόχο να ψηφίσουμε στην Επιτροπή 3 Μαΐου και να περάσει το θέμα στην Ολομέλεια την 1η του Ιουνίου. Αυτό είναι το τρέχον χρονοδιάγραμμα. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Δεν ξέρω ποιος δεν έχει πάνω του την κάρτα. Εγώ δεν την έχω πάντως. Την ξέχασα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Μπορεί κάποιος να πάει να μου τη φέρει. Για να δούμε τι γίνεται με τις κάρτες, πόσοι τις έχουν και πόσοι δεν τις έχουν. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών για να οργανωθούμε προκειμένου να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Συνάδελφοι, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία με τις ηλεκτρονικές κάρτες. Παρακαλώ ψηφίστε ό,τι θέλετε για να ελέγξουμε ότι λειτουργούν οι κάρτες. Open the vote. Open the vote. Έναρξη ψηφοφορίας.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 Right, we want, we want, we want. Okay, right, right. We want a repeat test. Can you, can you open the? Επανάληψη. Έναρξη ψηφοφορίας νούμερο 2. Α, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε. Α, τώρα μπορείτε να ψηφίσετε. Ψήφισαν όλοι. It's not a real vote, it's a test vote. And when do we see the surplus? Okay, no surplus. We have Okay, right, and at the moment we... You haven't got your card. Δεν έχεις την κάρτα σου. Μπορείς να στείλεις να στη φέρουνε. Καλό γατό. If it crucial, deal with the αν ε, υπάρξει πρόβλημα θα το χειριστούμε αργότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον που να περισσεύει, οπότε μπορούμε να περάσουμε στη ψηφοφορία της έκθεσης Γκαρθία Μαγκάγιου. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τοπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τοπολογία 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 32 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροποποίηση τώρα για να αλλάξει το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει αν αναγκαίως είναι υπέρ κατά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 τι είπατε. Ομού για τις υπόλοιπες. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ομού μέχρι τέλους υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνονται όλες αυτές λοιπόν μέχρι το τέλος. Θα ψηφίσουμε για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ, κατά, αποχές, κάποιες αποχές εκεί, και ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα υπέρ κατά αποχές δύο ψήφοι εναντίον δύο αποχές εντάξει εσείς είσαστε υπέρ και δύο αποχές εντάξει εγκρίθηκε λοιπόν συγχαρητήρια προς τον εισηγητή <laughs> um, περνάμε τώρα και ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κάζα. Έχετε το κείμενο μπροστά, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Μια στιγμή. Ωραία. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Ωραία. Τροπολογία 4. Ναι. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Είχατε χρόνο όμως, έτσι. Λοιπόν, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η προφορική τροποποίηση τώρα του ΕΛΚ την έχετε στο έγγραφό σας. Όσοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ναι, σωστό. Συμβιβαστική τροπολογία για την 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός τροπολογίας 16-17 και της ε, Jury 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία στι τροπολογίες 19 και 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και ψηφίζουμε το κείμενο πως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον συντάκτη, εισηγητή. Τώρα θα πάμε στην ψήφιση της δικής μου γνωμοδότησης. Εντάξει. Ήδη είχαμε συμφωνήσει. Θα ψηφίσουμε ομού συνολικά επί των τροπολογιών. Όσοι είναι υπέρ αυτών. Κατά αποχές ομόφωνα εγκρίθηκαν. Συγχαρητήρια λοιπόν για σε μένα την ίδια. Right. Um- Πολύ καλά. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Μάλιστα, τέλος ψηφοφοριών εδώ. Και τώρα θα συνεχίσουμε, θα περάσουμε για να δω μια στιγμή. Πολύ καλά. Στο σημείο 12 έχουμε τις τροπολογίες που θα εξετάσουμε όσον αφορά την, ε, τις ε, εγγυήσεις προς το κοινό και τις ε, απαιτήσει για τη διαφάνεια, τροποποίηση οδηγιών κτλ. Λοιπόν, ωραία. Θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι ότου επανέλθει ο εισηγητής. Εντάξει, ο Βολφ Κλίντς.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 Είχαμε μια πολύ καλή συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών εξετάζοντας ορισμένες εξαιρετικές συμβιβαστικές τροπολογίες και από ό,τι βλέπω έχουμε πολύ καλή συνένεση και αυτό είναι πολύ καλό γιατί βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ως Επιτροπή με όλες τις πολιτικές ομάδες και μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά από την συνάντηση που είχαμε μετά το γεύμα. <laughs> Επιστρέφει ο περιπλανόμενος. Ε, υπόθηκαν πίσω από την πλάτη σου ωραία πράγματα. Πού να άκουγες. Έχεις το λόγο, Βολφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Udo. ησυχία παρακαλώ. Ε. Ε, ε. Ο Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> στου σκιώδεις εισηγητές αλλά και στους άλλους συναδέλφους ευχαριστίες για τις ε, διάφορες τροπολογίες που κατατέθηκαν και ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές γιατί ήταν πρόθυμοι σε προσωπικέ συζητήσεις και επαφή μαζί μου να συζητήσουμε, να δούμε αυτές τις τροπολογίες. Πιστεύω ότι στην εκπόνηση συμβαστικών τροπολογιών <clears throat> προχωρήσαμε σχετικά πολύ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να αναφερθώ στα εξή θέματα. Δηλαδή, κύριοι επενδυτές, κατόφλια όσον αφορά καθορισμό του προνομιούχου επενδυτή, συμφωνούμε ότι στην Κασκάδε συμβαίνει το εξής. Ο εκδότης για το, περιεχόμενο του φυλαδίου είναι υπεύθυνο όταν ο ίδιος το εκπονεί ή όταν για τη χρήση δίνει εντολή σε τρίτους και αυτή η χρήση μπορεί να συνδέεται με κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Αν κάποιος διαμεσολαβητής χωρίς την άδεια χρησιμοποιεί αυτό το φυλάδιο, το ενημερωτικό αυτό, ή ίσως και το τροποποιεί, τότε είναι σαφές ότι είναι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση και είναι υπεύθυνο και για εκ των υστέρων συμπληρωθήσεις πληροφορίες, προσωπικά υπεύθυνο. Καταλήξαμε σύντομα σε συμφωνία, δεν πρέπει να εκπλήσει κανένα, είναι κανονικά κοινό νους αυτό που μας ε, ενέπνευσε. Τώρα για τους κυρίους επενδυτές θέλουμε και συμφωνούμε και από αυτού να διασφαλίσουμε ότι το φθινόπωρο εφέτος όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το πακέτο για αυτές τις επενδύσεις ε, θα το καταθέσει να μην καταλήξουμε σε διαφορετική αξιολόγηση και αντιμετώπιση αυτών που έχουμε εμείς για αυτά τα φυλάδια, για αυτές τις ενημερωτικέ ε, ε, εκδόσεις ε, και τις προτάσεις Επιτροπής. Απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει αυτά τα δύο έγγραφα να είναι συμβατά και συνεκτικά μεταξύ τους. Επί της αρχής υπάρχει συνένεση ότι είναι χρήσιμο να είναι ένα πιο σύντομο, πιο εύληπτο έγγραφο από αυτό που αυτή τη στιγμή αποτελεί τη σύνοψη, summary paper. <clears throat> Όσον αφορά τα, τις τιμές κατόφλια, μετά από ευρύτερη συζήτηση καταλήξαμε τελικά στο να πούμε ότι όσον αφορά τις επαφές και συζητήσεις ε, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θέλουμε να έχουμε 5 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2,5 εκατομμύρια ως τιμή. Θέλουμε να πάμε στα 5 εκατομμύρια, να δώσουμε ακριβώς ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν χρήση της κεφαλαιακής αγοράς χωρίς να υπάρχουν υπερβολικά περίπλοκα προσκόμματα και εμπόδια από πλευράς γραφειοκρατίας. Γι' αυτό <clears throat> για την εξαίρεση δεν θα είναι εξαίρεση μέχρι 2,5 αλλά μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι σκόπιμο νομίζω, έχει νόημα Όλοι θέλουμε, όχι μόνο κιόλα μετά την κρίση, όλοι θέλουμε συνολικά να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα εξαρτάται μόνο από τις τράπεζε, αλλά όλο και πιο πολύ να μπορούν να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται τις ε, υπηρεσίες τη ε, αγορά κεφαλαίων. Ο προσοντούχος επενδυτής που σε αυτή την ε, οδηγία αναφέρεται, πιστεύουμε ότι θα πρέπει επαρκώς να καθορίζεται και θα πρέπει αυτός ο ορισμός ε, να είναι κάτι με το οποίο θα συμμορφωνόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε τροποποίηση. Συμφωνούμε όμως ότι οι επενδυτές από πλευρά τους θα πρέπει αυτό το καθεστώς ενός προνομιούχου ή προσοντούχου επενδυτή να, ε, το, ε, να μπορούν να διαφοροποιηθούν και ίσως και ως μη επαγγελματίας επενδυτής να μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιες συναλλαγές και πιστεύουμε ότι δεν είναι πλέον αναγκαίο να έχουμε ένα ξεχωριστό μητρό. Ξέρουμε ότι εδώ εν μέρει στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για αυτό το θέμα, όπως π.χ. στην Ιταλία για την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεχωριστό μητρό, αλλά με την ερώτηση ποια ήταν η πείρα με αυτό το μητρό εκεί, έπρεπε να διαπιστώσουμε ότι ένα τέτοιο μητρό δεν υπήρχε καν εκεί. Όσον αφορά τις, ε, τα δικαιώματα έκδοσης, εμείς θα έπρεπε, και αυτό οι τελευταίες συζητήσεις με τους κοιόδης εισηγητές το κατέδειξαν, θα έπρεπε να διαφοροποιούμαστε σε σχέση με τις νέες ε, μετοχές και bonds ομολόγα. Ε, και εδώ τι συμβαίνει, θα πρέπει με αυτή τη διαφοροποίηση, για να υπάρξει αυτή τη διαφοροποίηση, μια τροπολογία του συναδέλφου θέλουμε να την λάβουμε υπόψη και να ενταχθεί ότι η διευκόλυνση όσον αφορά τέτοια δικαιώματα έκδοσης ε, θα πρέπει και για αυτά τα, για αυτά τα χρεόγραφα να λαμβάνονται υπόψη. Είχαμε και αρκετά μακρές συζητήσεις όσον αφορά τη διάρκεια ισχύω αυτού του φυλαδίου. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να παραταθεί η διάρκεια αυτή. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο μάλλον επιφυλάξεις έχει για κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά το θεώρησα πολύ μεγάλο προτέρημα, διότι στο βασικό φυλάδιο, στο φυλάδιο που επανειλημμένα χρησιμοποιείται για διάφορες εκδόσεις ε, ομολόγων και μάλιστα για μια σειρά μηνών ή και ετών ένα τέτοιο βασικό φυλάδιο πρέπει να έχει διάρκεια 36 μηνών. Θα πρέπει να θεωρείται ενισχύ για 36 μήνες. Συμφωνήσαμε τώρα με πραγματιστική προσέγγιση να αφήσουμε το φυλάδιο στα 12, στους 12 μήνες και το βασικό φυλάδιο να παραταθεί σε 36. Τώρα, εν τέλει, ένα θέμα στο οποίο ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο για να οριμάσει, αλλά μέχρι την ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα πρέπει να έχει αποσαφινιστεί οπωσδήποτε. Αυτό είναι η εισαγωγή ή η λήψη υπόψη MTFs, δηλαδή ε, Multilateral Trading Facilities, πολυμερείς ε, διευκολύνσεις εμπορίου. Θα τις αντιμετωπίσουμε όπως τις ε, ρυθμιζόμενες αγορές ή μήπως θα λάβουμε υπόψη ότι πρέπει άλλες προϋποθέσεις να ισχύουν εδώ. Άκουσα ότι πολλές, πολλά MTFs εθελοντικά, εθελούσια εντάσσονται στους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και θέλουν να εντάσσονται σε αυτούς όπως οι αντίστοιχες αγορές. διερωτώ με όμως αν επίσημα ε, θα έπρεπε να δοθεί ένα τέτοιο καταστατικό ή όχι. Εφόσον δεν το κάνουν αυτό επίσημα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν τους δίνουμε τα ίδια προνόμια αν, παρότι δεν εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο προστασίας. Μετά η αύξηση των κατοφλίων όσον αφορά τις εξαιρέσεις για το φυλάδιο, για τις κατατμήσεις. Τώρα αυτή τη στιγμή 50.000 ευρώ είναι η κατάσταση η προβλεπόμενη ως κατόφλι. Το αν θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό ως 50.000 ευρώ έχει, ή να το τροποποιήσουμε ως τιμή έχει διαφορετική απήχηση. Εμείς στο τέλος, νομίζω, τελικά, έτσι τουλάχιστον κατανόησα εγώ, με κάθε προσοχή και επιφύλαξη το λέω αυτό, γιατί ίσως ε, μπορεί μετά να μην έχει κατανοηθεί σωστά και να έχει αλλάξει αυτό, ότι στα 100.000 υπήρξε συμφωνία. Υπήρξαν ε, προτάσεις να πάμε μέχρι τα 250.000 ευρώ. Νομίζω 100.000 θα ήταν εντάξει ως τιμή. Αν, διότι ένας μέσος επενδυτής, ε, ιδιώτης, δεν θα δώσει παραπάνω από 50.000 ευρώ. Συμβαίνει καμιά φορά, αλλά είναι εξαίρεση για, ε, ως τάση. Και θα έπρεπε εδώ μια ρύθμιση τέτοιου είδους να μην την καθορίσουμε με ατομικές ε, περιπτώσεις ή εξαιρέσεις που δεν είναι ο κανόνας και δεν είναι το πιο σκόπιμο. Και γι' αυτό θα έλεγα εδώ αν θεωρούμε και συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια αλλαγή στο μέγεθος ή στην τάξη μεγέθους σε μεγαλύτερη τιμή, ε, τότε να δούμε την ε, επανεκπώνηση, την επανεξέταση ε, της ε, ρύθμισης αυτής. Αυτά για αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι συμφωνήσαμε στα κυριότερα σημεία. Το μόνο το οποίο απομένει και εκκρεμεί σημείο είναι πότε και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις Multilateral Trading Facilities, MTF, θα θεωρούνται ως ισότιμες ε, με ε, τις αγορές που θα έχουν ε, ρυθμιστεί. Θα έλεγα να μην το κάνουμε καλύτερα αυτό, να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Και εδώ να ελπίζουμε ότι με την επανεξέταση ή επαναδιατύπωση που μπορεί να υπάρξει όσον αφορά διάφορες οδηγίες, είτε είναι fit Market Abuse και τα για την ενασχόληση με αυτό το θέμα, να το ξαναδούμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει αυτό το σημείο θα πρέπει να το ψηφίσουμε αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Ευχαριστώ. Um, Προσπαθώ να δω ποιος θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Διόγκο. Yes. Ζητήσατε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ πολύ γοργά, θα έλεγα σύντομα, θα ήθελα να ευχαριστήσω μόνο τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε τον κύριο Βολφ Κλίντς και για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να επιτευχθούν συμβιβασμοί σε σχέση με διάφορα θέματα. Είναι μια οδός, μια πορεία που στέφεται με επιτυχία για τη διευθέτηση αυτών των θεμάτων. Στη συνεδρία συνάντηση που είχαμε ήταν καλή η συνάντηση και σε σχέση με τα όσα έγιναν από τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για αυτά τα ζητήματα. Θα θέλω επίσης να ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που έγιναν από διάφορους συναδέφους της ομάδας μου, καταθέτοντας ένα σύνολο τροπολογιών και αυτές εξετάστηκαν ως βάσεις ε, για κάποιο συμβιβασμό. Το τελικό μήνυμα λοιπόν για αυτό το θέμα θα έλεγα ότι υπάρχει ελπίδα να μπορέσουν όλα να λειτουργήσουν καλά μέχρι να έρθει η ώρα να ψηφίσουμε και να διευθετηθεί το θέμα. Κάθριν Στάιλα. Eh. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Σήμερα οι εισηγητές μας πρότειναν πολύ καλούς συμβιβασμούς που πολλοί από εμά θεωρούμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την προσέγγιση και το βασικό έγγραφο και το να μην προτιδικάζουμε τα αποτέλεσμα των προβασιλιστικών εργασιών στις συμβαστικές CD και E λατινικό. Για την H λατινικό έχουμε δουλειά να κάνουμε ακόμα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Για τα MTF, ξέρω ποια είναι η προσέγγιση του εισηγητή, χρειάζεται σαφήνεια και ελπίζω να τα καταφέρουμε συμφωνήσαμε συνεδρίαση για το κατόφλιο 50.000. Κάτι υπόθηκε για 100.000, είναι 50.000. Ε, ναι, βλέπω ότι συμφωνείτε, σηκώντε το δάχτυλό σας, μάλιστα, τον αντίχειρά σας. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας, Δόκτωρ Κλίντσον. Και μακάρι και στο μέλλον οι εργασίες αυτής της Επιτροπής να διεξαχθούν με τέτοιο τρόπο ένταξη, συμπερίληψη όπως ε, διεξάγατε και στις εργασίες. Η Πρόεδρος. Άλλο τι αγορεύει βούλεται. Πίτερ. Ο Βόλφ έδωσε σωστή εικόνα. Το κατάλαβε. Θα ήξερα ποια είναι η απόψη τους να ξέρω στα ευρύτερα θέματα. Λοιπόν, όσον αφορά τις τα φυλάδια, όταν συζητήσαμε τα φυλάδια, όταν ήταν ο Chris Χουνερ στην Επιτροπή, Chris συζητήσαμε εκτενώς πώς θα χρησιμοποιούσαν αυτού του είδους τα φυλάδια, αυτά τα διαβατήρια. Επιτρέπει η αντιμετώπιση παρόμοια πάλες οδηγίες. Είναι σοβαρή αυτή η αρχή και ελπίζω να το εγκρίνεις. Αν οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να χρησιμοποιήσουν τις κεφαλουχικές αγορές, να χρησιμοποιήσουν τους πόρους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή την αρχή. Χαίρομαι που το ακολουθείς αυτό και το λαμβάνεις υπόψη και το υπογραμμίζεις. Είναι η σωστή προσέγγιση. Συμφωνώ και όλοι συμφώνησαν με το θέμα MTF και Κάθριν. Δεν θέλουμε κανόνες περί συγκεντρώσεως για τη διαδικασία, δεν θέλουμε να εμφανιστούν μονοπόλια όπου μόνο κάποια χρηματιστήρια θα μπορούν να κινηθούν Ξέρουμε ότι αυτό δημιουργεί διαφορές και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ε, ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια κεφάλαια θα απαιτηθούν. Χρειάζεται συνένεση λοιπόν στην Επιτροπή επ' αυτού. Είναι ζωτική σημασία. Αν πετύχουμε τη συνένεση θα μας βοηθήσει και σε άλλες εκθέσεις. Θα πρέπει να διατηρήσουμε συνέπεια και συνέχεια αργότερα. Κυρίως μετά όταν μιλήσουμε για την AIFM. Άλλος, ο Βόλφ έχει το λόγο, Συγητής εκ νέου. Πώς δεν έχω να προσθέσω πολλά για τα σχόλια. Ελπίζω ότι γοργά θα καταφέρουμε τα τελευταία ένα-δύο σημεία που εκκρεμούν να τα διευκρινίσουμε ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Okay, Καλώς. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, 23 Μαρτίου, και έχουμε σαν στόχο την σύνοδο του Μαΐου, την Ολομέλεια του Μαΐου. Πάμε τώρα στο AIFM. Προχωρήσαμε πιο γρήγορα και χάσαμε και τον εισηγητή. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών περίπου, ούτως ώστε να εντοπιστεί ο εισηγητής και να προσέλθει. Ευχαριστώ.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 Okay, uh, Καλώς συγκεντρωθήκαμε όλοι εκ νέου. Αρκετά χρήσιμο το διάλειμμα, διότι καθόμουν στην καρέκλα επί διήμερων, χωρίς ανάπαυση μέχρι τώρα, οπότε ξετίμησα τα μάλα το διάλειμμα, παρόλο που ίσως μερικοί από εσά να μην το χρειαστήκατε. Έχουμε προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα, αλλά όπως γνωρίζετε αυτά τα χρονοδιάγραμματα είναι απλώς ενδεικτικά, οπότε πηγαίνουμε τώρα στη συζήτηση των τροπολογιών της οδηγίας για εναλλακτικά ε, για τους διαχειριστές για των ε, εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων θα δώσω το λόγο στον εισηγητή Ζων Πολ Γκουζές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τους ειδικού του περιβάλλοντος διότι του όγκου χάρτου που ετυπώθη αλλά ο κανονισμός του Κοινοβουλίου είναι τέτοιος που επιβάλλει οι τροπολογίες να παράγονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες που συζήτησε. Και όπως δεν ήσασταν τσιγκούνιδες όσον αφορά τροπολογίες όλοι σας, καταλήξαμε σε εντυπωσιακό πακέτο εγγράφων. Ας περάσουμε στο θέμα όμως. Εχθές το Συμβούλιο, ΕΚΟΦΗΝ, αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση επί της οδηγίας IFM που έπρεπε να λάβει η χώρα και για την οποία η Ισπανική Προεδρία είχε προτείνει ε, κάποιους συμβιβασμούς. Όταν έλαβα γνώση της αποφάσεως δεν το θεώρησα κάτι δραματικό. Γνώριζα ότι υπήρχε πολιτικό πρόβλημα όσον αφορά τις τρίτες χώρες το καθεστώς που θα επικρατούσε και η εγγύητης των Βρετανικών εκλογών μπορούσε να οδηγήσει, στο, να οδηγήσει τον Βρετανό Πρωθυπουργό να μην θέλει να λάβει μια απόφαση σε αυτό το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ διότι σύμφωνα σε δείξεις που μου δόθηκαν η Μεγάλη Βρετανία δεν είχε ε, μειοψηφία που μπορούσε να μπλοκάρει τις εργασίες. Δεν θα είναι από μακρύ ημερομηνία η επόμενη. Θα είναι ευκαιρία τότε η Ισπανική Προεδρία να ρυθμίσει περαιτέρω διαπραγματεύσει και να παρουσιάσει ένα συμβιβασμό στα κράτη-μέλη, συμβιβασμό που θα μπορούσε να υποστηριχθεί από όλου. Όσον αφορά το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι αυτή η αναβολή λήψος αποφάσεω ή τοποθετήσεω δεν θα πρέπει να διαταράξει το δικό μα ε, χρονοδιάγραμμα. Λέω δεν θα έπρεπε να το διαταράξει σημαντικά αν επρόκειτο απλώς να εκμεταλλευτούμε αυτό το συμπληρωματικό χρονικό διάστημα για να αναβάλουμε λίγο την ψηφοφορία ώστε ο φόρτος εργασίας μας να μειωθεί αυτό δεν θα ήταν και τόσο αρνητικό κατά την άποψή μου όμως δεν τίθεται θέμα θεωρώ να περιμένουμε μια θέση του Συμβουλίου πριν να τοποθετηθούμε εμείς και εξηγούμε στα δύο χαρτοφυλάκια που πρέπει να συζητήσω τα σημαντικά και που εξέτασα την, υπηρεσία, την οδηγία υπηρεσιών πληρωμών και τον κανονισμό για ε, τους διαφόρους αρμόδιους φορείς η, τοποθετήθηκε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τοποθετηθεί το Συμβούλιο στην προηγούμενη θητεία. Όσον αφορά τι υπηρεσίε πληρωμών, αυτή την οδηγία, αυτό ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Ψηφίσαμε στι 12 Σεπτεμβρίου, διαφορά του 2006, και το Συμβούλιο συμφώνησε τον Μάρτιο 2007 και τελικά ψηφίσαμε στην Ολομέλεια ένα συμβιβασμό στην πρώτη ανάγνωση τον Απρίλιο του 2007. Το ίδιο και για τους φορείς βαθμολόγησης ε, καταλήξαμε στην πρώτη ανάγνωση σε συμφωνία. Αυτά λοιπόν ήταν δύσκολα θέματα και ευαίσθητα. Το ότι εμείς τοποθετηθούμε θα πριν από το Συμβούλιο είναι ένα πλεονέκτημα διαπραγματευτικό. Και είναι καλό παράδειγμα για το Συμβούλιο όταν εργαζόμαστε καλά. Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να αλλάξουμε την αρχή αυτή, να ψηφίσουμε σύντομα με άλλα λόγια την έκθεση. Αντίθετα, ενδεχομένως, αν η ψηφοφορία στην Ολομέλεια αλλάξει η ημερομηνία, μπορεί να αλλάξει αν δούμε τη στιγμή θα τοποθετηθεί το Συμβούλιο ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για μια επικοδομητική και ικανοποιητική διαπραγμάτευση. Αυτά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα νομίζω ότι κανείς δεν θα κατανοούσε ούτε μεγάλο μέρος της κοινή γνώμης δεν θα καταλάβαινε μετά από αυτά που υπόθηκαν στου αρχικούς κρατών κυβερνήσεων και στους G20 αν εμείς σταματούσαμε όσον αφορά την οδηγία. Αυτό θα βόλευε εκείνος που είναι αντίθετοι τη οδηγία, αλλά ο εισηγητής ε, θα επλήγεται και το κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε να επιμείνουμε. Ε, και ακούσαμε αυτά που είπε και ο Επίτροπο το πρωί στην ε, συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εμεί θέλουμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά τη δουλειά που έγινε μετά από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, εγώ δεσμεύτηκα ούτω ώστε συμβιβαστικέ τροπολογίε να προταθούν πριν αυτή τη συνεδρίαση. Υπευλήθησαν στου Σκιώδη καταρχά, με του οποίου συναντήθηκα προχθέ και σε όλου του συναδέλφου που πρέπει να τι έχουν τι πρώτε συμβιβαστικέ Τώρα, βέβαια δεν υπήρχε πολύ χρόνο σου μεταξύ υποβολής των εγγράφων και τη συζητήσεω στην Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο όγκος των τροπολογιών που προτάθηκαν, ο περίπλοκος χαρακτήρας του θέματος, το θέμα ότι δεν είχαμε τις τροπολογίες που υπευλήθησαν παρά τις εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία, όλα αυτά μας δείχνουν ότι μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Έτσι δε μάλλον, διότι προσπαθήσαμε να ετοιμάσουμε συμβαστικέ τροπολογίε, όπω έλεγα, επί των πιο σημαντικών σημείων. Η συζήτηση με του Κιώδη ξεκίνησε, έλαβε χώρα. Δεν αναπόκειται σε μένα να πω ποια είναι η θέση των διαφόρων. Θα πω απλώς ότι πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλό συμβιβασμό στο Κοινοβούλιο και αυτό είναι πιο αναγκαίο τώρα από ότι αν δεν είχαμε έναν ευρέως αποδεκτό συμβιβασμό αν δεν είχαμε αυτόν τον ε, αποδεκτό συμβασμό θα είχαμε λιγότερα περιθώρια διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Και αν τυχόν ε, δείχναμε ότι είμαστε πολύ σκληροί αυτά τα αιτήματα, θα υπήρχε ο κίνδυνο να μην καταλήγαμε σε κάποια συμφωνία και να παίξουμε το παιχνίδι εκείνων που δεν θέλουν αυτή τη ρύθμιση, που είναι ε, κεφαλαιόδου σημασία και αναγκαιότητα. Εγώ προτιμώ να ακούσω τα σχόλια των διαφόρων και θα είμαι λακωνικό όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, το scope, Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε συμφωνία επί της βάσης των προτάσεων, δηλαδή να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα ταμεία που δεν πέτυχαν μπαίνουν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή οδηγία, αλλά με ελαφρύνσεις για εκείνους που δεν δικαιολογείται να υπόκεινται σε μια πάρα πολύ αυστηρή ρύθμιση. Για να δώσουμε κάποια ουσία σε αυτή την προσέγγιση, ε, προτείνω να τονίσουμε την αρχή της αναλογικότητας αλλά να μην περιοριστούμε σε αυτή τη δήλωση και υπογράμμιση. Εγώ προτείνω σε ένα παράρτημα να εμφανίσουμε τα είδη ταμείων, τα χαρακτηριστικά τους εκείνων που θα τύχουν ελάφρυνσης των τυπικών διαδικασιών και αυτό να είναι σαφές διευκρινίζοντας τις διάφορες διαδικασίες από τις οποίες θα απαλλαχθούν Επ' αυτής της βάσης μπορούμε ταυτόχρονα να ικανοποιήσουμε και εκείνους που επιθυμούν να μην ε, αυξήσουμε τα γραφειοκρατικά, τι εκλογικέ διαδικασίε και να σεβαστούμε τι γενικέ αρχέ σύμφωνα με τι οποίε κάθε χρηματοστατική δραστηριότητα θα πρέπει να ρυθμίζεται και να ελέγχεται. Προτείνω, αλλά συζητείται ακόμα αυτό, να επανεισαχθεί το κατόφλιο όχι για την ε, απαλλαγή από την οδηγία για τις εξαιρέσεις αλλά για να λάβουμε υπόψη τα ταμεία που είναι μικρού μεγέθους, μικρής κλίμακας, ώστε η ρύθμιση να προσαρμόζεται κατά αναλογία. Τόσο αφορά το private equity, και αυτό κατά την άποψή μου ελαφρύνεται σημαντικά για να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα αυτής της δραστηριότητας και του, να λάβουμε υπόψη και το κίνδυνο που αντιμετωπίζει. Να πω ότι ο στόχος της ρυθμίσεως είναι η μεγαλύτερη νομική ασφάλεια εποπτεία, ρύθμιση και δεν πρόκειται απλώς για την πρόληψη του συστημικού κινδύνου. Η κρίση μπορεί να προέλθει από άλλες πηγές, πέραν του συστημικού κινδύνου. Το ότι λέμε ότι εμείς δεν, ε, δεν υποστηρίζουμε συστημικό κίνδυνο δεν είναι επαρκές ε, ε, επιχείρημα για να απαλλαγούμε από τις γενικές υποχρεώσεις ρύθμισης και εποπτείας. Όσον αφορά το πλέον ευαίσθητο θέμα των τρίτων χωρών, επ' αυτού το Συμβούλιο έχει κολλήσει. Από όταν υπέβαλα την εκθέση μου άλλαξα κάποιες θέσεις. Είχα πει ότι η αρχική μου πρόταση ήταν, προ... ήταν προτάσεις αναμονής. Να δω πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες μεταξύ μας. Η που κάνω σήμερα, η πρόταση που κάνω σήμερα είναι μια πρόταση που υποστηρίζει τις ιδιωτικές ε, τοποθετή επενδύσεις για μια ε, προσωρινή περίοδο πενταετή επιτρέποντας προπτική κάποιας ρύθμισης που μπορεί να ασχίσει και για τρίτες χώρες και θα επέτρεπε σε διάφορους χειριστές πόρων εκτός ταμείων εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αφαιρηθούν από τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Η μία είναι η αναγνώριση μιας ισοτιμίας ισοδυναμία. Τα κράτη-μέλη που είναι επιφυλακτικά στον αφορά ισοδυναμία δεν διαμαρτύρονται τόσο για την ενεργή φάση της εμπορευματοποίησης όσον αφορά τι θα συνέβαινε όταν σε μια τρίτη χώρα θα για κάποια δικαστική υπόθεση και η νομολογία τη τρίτη χώρα σε περίπτωση χρεοκοπία δεν θα είχε την ίδια στάση όπω αυτή που θα είχε ένα Ευρωπαίο δικαστή. Είναι ένα επιχείρημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και γι' αυτό το λόγο Πιστεύω ότι αυστηρά κριτήρια σημαντικά και σαφή θα πρέπει να τίθεται όσον αφορά την αναγνώση της ισοδυναμίας. Αυτό προϋποθέτει ότι σαφώς θα πούμε ποια θα είναι η αρχή ή οι αρχές που δίνονται να παρέμβουν στην παροχή της ισοδυναμίας γνωρίζετε ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει φόβος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέψτε να το πω, δεν θα ήταν αρκετά στέρεη για να αντισταθεί σε αιτήματα ισοδυναμίας που δεν θα δικαιολογούνται. Θα ήθελα όμως παρόλα αυτά να προβώ σε κάποιο σχόλιο όσον αφορά αυτό το επιχείρημα των ξένων νομολογιών. Σήμερα στις περισσότερες χώρες ή σε πολλές χώρες οι ιδιωτικές επενδύσεις επιτρέπουν στους θεσμικούς επενδυτές να αγοράσουν πόρους εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να επενδύσουν σε ταμεία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή να αγοράσουν ε, ταμεία και πόρους που παρουσιάζονται από διαχειριστές πόρων που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τοποθετήσεις, με ενεργό μάρκετινγκ ή το παθητικό μάρκετινγκ που είναι υποκριτικό. Δηλαδή, ε, ε, κάπου ε, ο, ο θεσμικός επενδυτής λέει ότι υπάρχει κάποιος ενδιαφέρον πόρο σε μια τρίτη χώρα και θα πάμε να αγοράσουμε. Είναι υποκριτικό σύστημα αυτό που θα πρέπει να καλυφθεί. Τούτων λεχθέντων, σε αυτά τα συστήματα, ο κίνδυνος που καταγγείλουν αυτοί φοβούνται την ισοδυναμία υπάρχει. Όταν ένας ε, θεσμικός επενδυτής Γάλλος, Φερρυπίν, αγοράζει ένα ταμείο στις, στα νησιά Καϊμό, δεν το παγορεύει κανείς, αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο αν υπάρχει δυσκολία. Ο, ο δικαστής των ίσων Καϊμάν θα κρίνει και θα κρίνει σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Είναι φόβοι ε, που θα πρέπει να σχετικοποιηθούν όμως. Προτείνω στη μεταβατική αυτή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι ιδιωτικέ επενδύσει υπάρχουν ω τώρα, ισχύουν ω τώρα, επιδιώκοντα αυτή την περίοδο να βρούμε ενδεχόμενη δυνατότητα ισοδυναμία με κάποιε χώρε, υπό αυστηρέ συνθήκες, το είπε και επίτροπο, και στι δύο περιπτώσει, είτε στο τέλο αυτής τη προσπάθεια εξευρέσεως ισοδυναμία κάποια τρίτη χώρα θεωρείται σαν ισοδύναμη και τι αυτή η περιπτώση οι χειριστές που, που βρίσκονται σε ισότιμη θέση με αυτού που βρίσκονται εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αυτή τη χώρα, ή δεν αναγνωρίζει τη ισοδυναμία και εκεί υπάρχουν δύο λύσει. Είτε μια ριζική λύση όπου τα ταμεία αυτής της χώρας ή που εμπορευματοποιούνται από τους διαχειριστές που είναι σε αυτή την χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαγορεύονται, απαγορεύεται η εμπορευματοποίησή τους εντός Ευρώπης. Αυτή αυτη τη χωρα η που εμπορευματοποιουνται απο του διαχειριστε που ειναι σε αυτη την χωρα εκτο ευρωπαικη ενωσεω απαγορευονται απαγορευεται Η εμπορευματοποιηση του εντο ευρωπη αυτη είναι ότι ιδιωτικέ επενδύσεις επενδυσει υπαρχουν για αυτές τις χώρες σε εθνικό επίπεδο που τις επιτρέπει. Μπορεί να υπάρξει και τρίτο ενδεχόμενο, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί 28 ε, 8 καθεστώ ιδιωτικών επενδύσεων που επιτρέπει να θεσπιστούν του εφαρμοστέου κανόνε για την εμπορευματοποίηση όταν τα υπόρρια αυτή, τα ταμεία αυτά ή οι χειριστέ του, διαχειριστέ δεν βρίσκονται εντό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Κάποια τροφή προσκέψη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια απόφαση εντό τη Επιτροπή μα. Από την πλευρά μου εγώ είμαι ανοιχτό προφανώς να ακούσω συστάσεις ε, που ε, ήδη αναφέρθηκαν από τους συντονιστές. Όσον αφορά το, τη συνέπεια, το, το αποτέλεσμα χρήσεως μοχλού, το σύστημα μόχλευση, το αποτέλεσμα μόχλευση, αυτό είναι και θέμα του διαχειριστού, αλλά η εποπτική αρχή θα πρέπει να μπορεί να το ελέγξει. Οι εθνικέ αρχέ τη στιγμή τη παρουσίαση του, του φυλαδίου ή του ημεριστικού σημειώματο που θα πρέπει να περιέχει σαφή στοιχεία όσον αφορά το ε, φαινόμενο μόχλευση που χρησιμοποιεί ο διαχειριστή του ταμείου και η εθνική αρχή κατά τη διάρκεια τη ζωή του Ταμείου θα πρέπει να επαληθεύσει κατά πόσο διαχειριστή σέβεται την πολιτική που υποανακοίνωση Και για να αποφευχθεί ο κίνδυνο που θα μπορούσε να απορρεύσει από μια υπερβολή όσον αφορά το φαινόμενο μόχλευση, η, η Ευρωπαϊκή Αρχή θα πρέπει κάθε φορά που θεωρεί ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η χρηματοπιστωτική ασφάλεια υπονομεύεται, διακινδυνεύει, να προβλέπεται η δυνατότητα να καθορίσει αυτή περιοριστικούς κανόνες όσον αφορά το φαινόμενο ομόχλευσης είτε εν γέννη είτε ενδεχομένως έναντι συγκεκριμένου διαχειριστού αν υπάρχουν αρνητικές ε, πληροφορίες που δίδονται σχετικά με αυτόν από τις εθνικές ε, αρχές. Αυτά όσον αφορά το φαινόμενο, το ποτέσμα μόχλευσης. Υπάρχουν και άλλα θέματα εκκρεμή, ε, θα τα αναφέρουν αυτά οι συνάδελφοι, κυρίως αυτό που κατευθύνεται, ποιο, ποια είναι η ευθύνη του καταθέτου να καθορίσει τη ευθύνη, να μην είναι μια ευθύνη που καλύπτει τα πάντα, αλλά να μην είναι ευθύνη σαφώ καθορισμένη, αποφεύγοντα όμω, ο καταθέτης να μπορεί να οργανώνει ο ίδιος ποιε είναι οι ευθύνε του, όπως τις εννοεί αυτός, μεταφέροντας, μετακυλώντα την ευθύνη του σε κάποιου άλλου. Στι περιπτώσει όπου η ευθύνη του καταθέτου ε, κινητοποιείται θα πρέπει να καθορίζεται σαφώ όμω, δύο περιπτώσει είναι όπου εκεί όπου ο νόμος της χώρας που είναι η κατέθεση θα πρέπει να προβλέπει να ε, παραμένει εκεί ο καταθέτης και σε περίπτωση που υπάρχει μια συμβατική απόφαση που μπορεί ε, να, κατά που μπορούν να προσφύγουν οι επενδυτές που πρέπει να το ξέρουν πριν λειτουργήσει το ε, ταμείο. Και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η περίπτωση του reuse, της εκ νέου χρήσης. Μετά τις συζητήσεις που είχα, είδαμε ότι μορφώνεται μια πλειοψηφία όσον αφορά την αμοιβή που θα πρέπει να αρμόζεται ε, επί τη βάση των αμοιβών των τραπεζών. Δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση. Ο κανονισμός του, περί φαινομένου μόχλευσης θα πρέπει να απαγορεύεται το φαινόμενο μόχλευσης όταν εκείνος που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τρόπο κίνησης δεν έχει κανένα δικαίωμα όσον αφορά τα αξιόγραφα και τα αγαθά τα οποία τη δεδομένη στιγμή θα πρέπει να παραδώσει. Αυτές είναι κάποιες προτάσεις, αλλά εγώ επιμένω εάν θέλουμε να αναβάλουμε κάποιες μέρες να δώσουμε κάποιο χρόνο παραπάνω για να σκεφτούμε το θέμα, αν αναβάλουμε την απόφασή μας για την ψηφοφορία, αυτή η απόφαση θα πρέπει όμως να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Ρόμπερτ Γκέμπερς, παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Καταρχάς να συγχάρω τον Σαν ε, Κοζέσια για όλη τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και για τον τρόπο που έχει χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις Νομίζω ότι αυτό προϊονίζει καλά αποτελέσματα και να πω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να καταλήξει σε μία απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία για αυτή την πρόταση. Γιατί μόνο αν έχουμε μεγάλη πλειοψηφία θα μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι στο Συμβούλιο. Όπως και ο Ζαν Πολ χαίρομαι πολύ που η Ισπανική Προεδρία δεν επέμεινε τελικά στο να εξεταστεί το θέμα στο χθεσινό ΕΚΟΦΗΝ. Γιατί έτσι έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε και με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή. Μας δίνει λοιπόν δυνατότητες μόχλευσης μεγαλύτερες για να μείνουμε στο κλίμα. Βεβαίως, Θεωρώ ότι η προσέγγιση της Ισπανικής Προεδρίας δεν είναι η κατάλληλη. Νομίζω ότι προσπάθησε να κάνει υπερβολικές ε, υπερβολικούς συμβιβασμούς να δώσει πολλές ε, επιλογές στα εθνικά κράτη κάτι όμως που διακινδυνεύει τη θέση της εσωτερικής αγοράς αλλά και ορισμένων βασικών πολιτικών. Νομίζω ότι η πολιτική της ήταν κακή και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς τη δημιουργία δηλαδή μιας πραγματικά εσωτερικής αγοράς και για τα εναλλακτικά κεφάλαια. Προφανώς ε, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη για όλες τις πάνω από 1600 τροπολογίες. Όμως, ένα πολύ ενδιαφέρον ήταν η τροπολογία 55 του Wolf Klintz που αναφέρει ότι η παρούσα οδηγία συμφωνεί με τον κανόνα που αναφέρθηκε στο Pittsburgh το 2009, σύμφωνα με το οποίο όλες οι αγορές, όλα τα προϊόντα, όλοι οι φορείς πρέπει να ρυθμίζονται σωστά. Θα ψηφίσω υπέρ αυτής της τροπολογίας που μας δείχνει τα βασικά. Διαπιστώνω όμως ότι πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν τροπολογίες που ζητούν εξαιρέσεις για διάφορα είδη κεφαλαίων, αλλάζοντας τα κατόφλια, επιτρέποντας στα μικρά κεφάλαια να διαφύγουν τις νομοθεσίες. Να πω ότι εγώ προσωπικά είμαι κατά αυτού του είδους των εξαιρέσεων. Είναι λάθος να λέμε ότι επειδή κάποιος είναι μικρός δεν δημιουργεί συστημικούς κινδύνους. Μας είπε ο Μάριο Ντράγκη ότι περίπου 50% των συναλλαγών στις, ε, εσωτε... στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές γίνονται μέσω των αναλλακτικών κεφαλαίων και ταμείων. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι και ο δικός τους ρόλος. Γι' αυτό θέλουμε να ρυθμίζονται σωστά. Γιατί ακόμη και οι μικροί μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε μεγάλες ζημιές. Τώρα όσον αφορά την κερδοσκοπία, για παράδειγμα στο πετρέλαιο. Ας δούμε το IMAX στη Νέα Υόρκη. τότε είχε αγοράσει κάποιος χίλια βαρέλια με 100 δολάρια το βαρέλι και αμέσως τα πούλησε χάνοντας χρήματα. Όμως με αυτή τη μία συναλλαγή δημιούργησε πρόβλημα για όλα τα υπόλοιπα hedge funds γιατί είδαν ότι το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό το σημαντικό ψυχολογικό φράγμα. Και αυτή μια συναλλαγή δημιούργησε πρόβλημα και άφησε τα σημάδια της σε όλη την παγκόσμια οικονομία. διαβάσαμε επιστολές που αφορούν άτομα που διαχειρίζονται κάποιες δεκάδες εκατομμύρια λίρες, στερλίνες ή ευρώ και άρα δεν μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες ζημιές. Κοιτάξτε, δεν θέλω να αμφισβητήσω τη χρησιμότητα αυτού του κλάδου. Όμως, σπάνια τα hedge funds λειτουργούν μεμονωμένα και ακόμη και η απόφαση ενός μικρού κεφαλαίου μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές. Είμαι λοιπόν υπέρ της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας και από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε δυνατότητες ελάφρυνσης ε, για κάποια κεφάλαια που βρίσκονται κάτω από ένα κατόφλι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε αυτό που ανέφερε ο Κλίντ στην τροπολογία του. Όλοι οι φορείς, όλες οι αγορές, όλα τα προϊόντα πρέπει να υπόκεινται σε καλές ρυθμίσεις και εγώ θα έλεγα και σε καλό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Παραμένουμε στους ισχυώδεις εισηγητές. Βολφ Κλίντς, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστίες πρώτα και έπαινο προς τον Ζαν Πολ Γκοζές που πραγματικά έκανε Ηράκλειο έργο εδώ. Έπρεπε να επιτελέσει Ηράκλειο έργο. Και έχει αντέξει και θέλουμε να τον υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο να ολοκληρώσει όσο καλύτερα γίνεται. με την άποψή του ότι εμείς στην Επιτροπή πρέπει πριν από το Συμβούλιο να ψηφίσουμε και να διευθετήσουμε. Σίγουρα λυθεύει. Αλλά δεν είμαι βέβαιος αν γι' αυτό στην πέμπτη ταχύτητα βιαστικά ή με την έκτη με εξατάχυτα αυτοκίνητα πρέπει να τρέξουμε αν πραγματικά πρέπει στις 12 Απριλίου να ψηφίσουμε και όχι κάποιες μέρες αργότερα. Το αφήνω ανοιχτό αυτό να το σκεφτούμε. Πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε αρκετό χρόνο ώστε επαρκώς να εξετάσουμε τα θέματα αυτά και να τα συζητήσουμε μεταξύ μας αν θέλουμε να έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία. Η τελική ψηφοφορία όμω στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει να γίνει πριν από το Συμβούλιο, χωρί αμφιβολία. Διότι χρειαζόμαστε εντολή ώστε να γίνει διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο από πλευρά μα και η θέση μα να είναι το δυνατόν καλύτερα διατυπωμένη στι διαβουλεύσεις. Υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν κέρια σημασία. Θα ήθελα να τα αναφέρω. Καταρχήν προ τον Ρομπέρ Γκέμπερτ. Από αυτά που ως τροπολογίες πρότεινα δεν έχω τίποτα να αποσύρω. Παρ' όλα αυτά, ένα σημείο θα ήθελα να συμπληρώσω ή να αποσαφηνίσω. Όταν εμεί συμφωνούμε και λέμε ότι στο σκόπ, στο εύρος, αυτό στο φάσμα, κάποια ταμεία πρέπει να εξαιρεθούν, επειδή αυστηρός σε εθνικό επίπεδο πολλούνται και ρυθμίζονται και επιτηρούνται, ε, τότε το αίτημά μου <clears throat> ανταποκρίνεται σε αυτό το γεγονός. Επιτηρούνται, ρυθμίζονται, ωστόσο όμως Μόνο, πώς είπατε, χωρίς μικρόφωνο. Εντάξει, έστω. Λοιπόν, κατά τούτο παραμένω στην αρχική μου διατύπωση, αλλά συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, το ότι ένα ειδικό ταμείο που μόνο από έναν πάροχο ε, υποβάλλεται και μόνο σε, ένα, σε μια χώρα ε, εντάσσεται και λειτουργεί να εξαιρείται. Φτάνω τώρα στο εύρος, στο φάσμα. Το συζητήσαμε ήδη αυτό. Ξέρει τις απόψεις μας ο κύριος Γκοζές Στη δική μου τροπολογία 1, πρώτον πρότεινα το πακέτο να επαναπεμφθεί και μια εξειδικευμένη οδηγία για hedge funds να ζητηθεί και μια περαιτέρω εξειδικευμένη για private equities. Για διάφορους λόγους δεν γίνεται αυτό, το γνωρίζω αυτό και έτσι δεν θα έχω πλειοψηφία στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. παρόλα αυτά ήθελα να διατυπώσω το αίτημα αυτό. Επειδή απλά το θεωρώ σωστό, έτσι. Γιατί το θεωρώ σωστό, γι' αυτό το ζήτης, το λέω. Εμείς εδώ πραγματικά έχουμε υπερβολικά ταμεία τα οποία τα εντάσσουμε και τα προσπαθούμε να τα καλύψουμε σε μια οδηγία. Θα ήταν για παράδειγμα πολύ καλύτερο <clears throat> τα state funds με users, με χρήστες να συνδυαστούν ξεχωριστά να... Ε, ε, αλλά τέλος πάντων μια ομάδα ε, παϊόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα διατύπωσε αυτά. Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα, δεν χρειάζεται εδώ να κολλήσουμε. Παρ' αυτά πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιοι καλοί λόγοι, κάποια ταμεία να εξαιρεθούν από αυτή την οδηγία. Πάντα υπό την προϋπόθεση ότι εθνικά θα προσφέρονται και θα απολούνται τα προϊόντα τους και θα ρυθμίζονται εθνικά ε, σαφώς και θα υποπτεύονται. Δεύτερο σημείο, τρίτα κράτη. Πραγματικά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Επανειλημμένα είπαμε ότι η Ευρώπη δεν θέλουμε να είναι χειρό, φρούριο. Δεν θέλουμε όμως να είναι ούτε και φυλακή η Ευρώπη. Ευρωπαίοι επενδυτέ να μην μπορούν ξαφνικά να επενδύουν σε θέματα σε πράγματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, συμφωνώ με τον Ζαν Πογκοζές, να βρούμε μια λύση εδώ που με τη βοήθεια κάποια μεταβατική περίοδου για τα ταμεία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δίνουν μια δυνατότητα σύγκληση να ε, καταδειχθεί ότι συγκλίνουν και έτσι να μπορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιούνται. Για μένα υπάρχει αυτό το ερώτημα που απομένει. Αν αυτό πράγματι συμβαίνει είτε η μεταβατική περίοδος θα είναι τρία ή πέντε χρόνια, θα το δούμε. Ε, τότε ένα ταμείο, θα έλεγα, που έχει έδρα στα νησιά Καϊμάν, θα μπορεί να δείξει ότι συγκλίνει για να μπορέσει να λειτουργήσει έτσι. Αλλά αυτά διαρκούν το χρόνο τους βέβαια. Και πέρα από αυτά πιστεύω εγώ ότι εμείς ως Ευρωβουλή στη διατύπωση των κριτηρίων που θα καθορίζουν αν υπάρχει δέσμευση όσον αφορά την σύγκληση. Δεν θέλω αυτό πλήρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαφεθεί, να πει μετά από κάμποσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ, κακό, πολύ δυστυχώ το διαπραγματευθήκαμε, αλλά 80% δεν έχουν σύγκληση από αυτού και δεν θα ξέρουμε αν θα είναι τα σωστά κριτήρια αυτά. Αυτό έγκαιρα θα πρέπει να πιέσουμε να εντάσσονται και να, είναι, να δεσμεύονται. Τώρα, για το αν τα κριτήρια θα είναι συνολικά και έτσι θα πρέπει να ενταχθούν εδώ, δεν το ξέρω, αλλά πρέπει τουλάχιστον να διεκδικήσουμε αυτό το δικαίωμα από πλευρά μα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιβεβαιωθεί ότι στην διατύπωση των κριτηρίων αυτών θα έχουμε λόγο να αρθρώσουμε ω Ευρωβουλή. Κατά πόσον αυτέ ε, οι ε, διατάξει θα ισχύουν, για ποια διάρκεια, πρέπει και αυτό να το ρυθμίσουμε αν έχουμε ένα καθεστώς ε, των 28, τότε φυσικά αυτό θα είναι, ας το πω έτσι, η κατάληξη. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, αν το Συμβούλιο εμείνει και επιμείνει και υπάρχουν κάποιοι στο Συμβούλιο και πούν ότι ένα ταμείο που βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ποδιαχειριστής του είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και αν συγκλίνει δεν θα έχει τέτοιο διαβατήριο, τέτοια ανάδεια λειτουργίας. Αυτό φυσικά είναι κάτι πολύ σκληρό. Αν συγκλίνει πιστεύω ότι σίγουρα θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο διαβατήριο, μια τέτοια άδεια. Αν δεν πάρει όμω τέτοιο διαβατήριο, πρέπει να έχει την δυνατότητα με βάση το καθεστώς αυτό να το χρησιμοποιήσει για να συναλλάσσεται στα κράτη-μέλη. Γιατί διαφορετικά θα είμαστε στεγανοί εμείς ως Ευρώπη. Δεν μπορεί να είναι αυτό το συμφέρον μας. Για παράδειγμα, ε, όσον αφορά συνταξιοδοτικά ταμεία και τέτοιες ε, δυνατότητες. Εδώ πρέπει να αποσαφνίσουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Εγώ θέλω να πετύχουμε ένα ταμείο που θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ο διαχειριστής θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα ταμείο που θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διαχειριστής εκτός Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής να μπορούν να συγκλίνουν για να λειτουργήσουν σε ένα ενίο πλαίσιο. Αυτό θα έλεγα μπορεί να γίνει ή θα έπρεπε να μπορεί να επιτευχθεί. Πέρα από αυτά έχω και ένα άλλο σημείο. Αφορά τη μόχλευση, το λεβίε, το, την δυνατότητα μοχλικής α, απόδοσης. Και πρέπει να ομολογήσω ήμουν εγώ ένθερμος υποστηρικτής του να ληφθεί υπόψη η μόχλευση ή από πλευρά ορισμού, ώστε η μοχλική απόδοση όχι μόνο μεταξύ hedge funds και private equities και τα λοιπά, να δούμε ότι είναι διαφορετική, αλλά ακόμα και στην ίδια κατηγορία υπάρχει διαφορετική απόδοση, διότι εξαρτάται ποιος όχι μόνο ποιο συντελεστή ενεργοποιούμε, αλλά ποια κατηγορία, σε ποια ε, ε, δρούμε. Η μία είναι ίσως αντιμετωπίζει περισσότερου κινδύνους από την άλλη, εγκυμονεί περισσότερου κινδύνους. Και να μην ξεχνάμε ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι τράπεζες. Διότι οι τράπεζες είναι εκείνε που πρέπει να ρυθμιστούν με αυστηρό πνεύμα και να πληρώσουν. Διότι οι τράπεζες για παράδειγμα, όταν χρηματοδοτούν τη συμμετοχή σε private equity με τόσο ποσοστό ξένου κεφαλαίου, αυτές οι τράπεζες είναι που δυσανάλογα χρησιμοποιούν υπερβολικά γενναιόδορες, ας το πω έτσι, δόσεις. Τώρα είναι πολύ χαμηλά βέβαια αυτές οι συναλλαγές, αλλά ξέρω ότι μια τράπεζα που ασχολείται για παράδειγμα σε σχέση με private equities και όταν πολλαπλά έχει χρήση ξένου κεφαλαίου ότι πάει υπερβολικά μακριά αυτή η δραστηριότητα. Αυτό μου θυμίζει την subprime χρηματοδότηση με συναλλαγές οι οποίες δεν είναι ε, φερέγγες. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν στην οδηγία για, τα, για τις τράπεζες Βασιλεία 3 ή 4 να εντάξουμε κάτι να υποχρεώνει τις τράπεζες σε σχέση με τα κεφάλαια που διαθέτουν να είναι συνετές και να χρησιμοποιούν ε, ε, την σύνεση στην στη διάθεση των ε, ε, χρημάτων. Να δούμε και τους private brokers, ε, τη διαφάνεια. 10-12 είναι παγκόσμια. Αυτοί ακριβώς πρέπει να μας πούν τι δίνουν ως ποσό σε ποιον, για ποια χρήση. Τότε θα υπάρχει διαφάνεια και τότε καταρχήν θα μπορεί ο κίνδυνος, τέλος πάντων όχι εμείς, οι επόπτες, οι επιτηρητές θα μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο ή τους κινδύνους και πιθανόν θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει και οι τράπεζες να καταλήξουν να είναι πιο συνετές, πιο λογικές στις δράσεις τους. Τελευταία παρατήρηση. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε ταμείο, είτε hedge funds, είτε private equities, σε εισαγωγικά πρέπει να τιμωρηθεί, να πληγεί από εμάς. Δεν είναι αυτό ο στόχος μας. Ε. Αλλά ένα πράγμα είναι σαφές. Τα hedge funds από εμά δεν μπορούν να αναμένουν συμπόνια όταν σε σχέση για παράδειγμα με το ευρώ και την ε, Ελλάδα κερδοσκοπούν έχω μηδενικό επίπεδο συμπόνιας και κατανόησης ε, για την δράση αυτή, για την τοποθέτησή τους. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Πασκάλ Καμβέ. Θα συμφωνήσω και εγώ με τα συγχαρητήρια που έχουν δοθεί για τον τρόπο που χειρίζεται τις συζητήσεις ο Ζαν Πολ Κοζέτς έχω λιγότερη εμπειρία από τους άλλους συναδέλφους πάντως ε, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να υπάρξει ψηφοφορία στο κοινοβούλιο πριν τη συζήτηση στο συμβούλιο. συμφωνώ λοιπόν με την πρόταση του Ζαν Πολ προκειμένου να κρατήσουμε μια ημερομηνία τον Απρίλιο. Τώρα, Έχουμε συζητήσει γενικά το θέμα, δεν θα επαναλάβω αυτή τη συζήτηση, απλά θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία της ανάλυσης όσον αφορά τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ο, καταρχάς όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ μας. Το σίγουρο είναι ότι αν θέλουμε να δώσουμε εξαιρέξεις σε κάποια κεφάλαια με βάση τη νομική τους υπόσταση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία κάποιο είδους ρήτρα έτσι ώστε αν χρησιμοποιηθεί αυτός ο τύπος κεφαλαίου προκειμένου να παρακαμφθεί η οδηγία θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα κάποιος να μπορέσει να αλλάξει το καθεστώς για το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Αν λοιπόν ε, η εξαίρεση αν λοιπόν ο συμβιβασμός μας θα προβλέπει εξαιρέσεις, θα ήθελα να υπάρξει μια τέτοια ρήτρα γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κίνδυνος επίσης να εξαιρεθούν πλήρως τα private equities με βάση τα κατόφλια των 150 εκατομμυρίων. Και βεβαίως αν ε, βάλουμε μία εξαίρεση της εξαίρεσης στο παράρτημα, ειδικά για τα private equities, μπορεί να καταλήψουμε στην πλήρη εξαίρεση των private equities, κάτι που νομίζω ότι δεν θέλει ο εισηγητής. Όσον αφορά τη μόχλευση τώρα, συμφωνώ με τον τρόπο που παρουσίασε τα πράγματα ο Σαν Πόλου δεν μίλησες για έκτακτες ε, συνθήκες και όντως οι πράσινοι δεν θέλουν να συμπεριληφθεί στο συμβιβασμό η έννοια των εξαιρετικών ε, ή έκτακτων συνθήκων. Νομίζω ότι αν το κάναμε αυτό τώρα όλοι θα λέγανε ότι είναι υπερβολικά αργά. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα πριν καταλήξουμε να αντιμετωπίζουμε έκτακτες συνθήκες. Όσον αφορά τώρα τρεις τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε το συμβιβασμό προς τον οποίο κατευθυνόμαστε, δηλαδή μεταβατική περίοδος και μετά ένα είδος διαβατηρίου και καθεστώτος καθαρά ευρωπαϊκού. Όμως, κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις. Υπήρχαν αντιρρήσεις για το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε αυτές τις αντιρρήσεις όσον αφορά τις αρχές επί της ισοτιμίας. Αν λοιπόν ο συμβιβασμός στον οποίο θα καταλήξουμε θα είναι μετά από τη μεταβατική περίοδο να συμπεριλάβουμε αυτή την αρχή της ισοτιμίας θα πρέπει να το κάνουμε με βάση τα πραγματικά στοιχεία. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα ήταν να υπάρχει αμοιβαιότητα στην αρχή της ισοτιμίας. Δηλαδή να ανοίγουμε την αγορά μόνο αν κάνει το ίδιο και η τρίτη χώρα. Επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε περιορισμό στο χρόνο της ισοτιμίας, δύο-τρία χρόνια κτλ. Θα μπορούσαμε επίσης να ζητήσουμε από την Κομισιόν να εξετάζει κάθε δύο-τρία χρόνια ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με την αρχή της ισοτιμίας. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες επιλογές και οι οποίες νομίζω ότι ανταποκρίνονται στους φόβους των κρατών μελών προκειμένου να μην μείνει η συμφωνία στα χαρτιά. Κάτι άλλο που μπορεί να συμπεριληφθεί είναι διασύνδεση της Κομισιόν με έναν άλλον οργανισμό που θα δίνει αυτές τις ισοτιμίες. Θα μπορούσε για παράδειγμα η Κομισιόν να ζητάει την γνωμοδότηση κάποιας τεχνικής, ας το πω έτσι, αρχής, η οποία θα καθοδηγεί τη συζήτηση και έτσι θα μπορεί και η Κομισιόν να βασίζεται στην γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΣΜΑ για να προχωρήσει σε κάποια απόφαση. Κάτι άλλο. Όσον αφορά το σεβασμό των κριτηρίων, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στην νομοθεσία της χώρας όπου βρίσκονται οι μάνατζερ, συνήθως οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και τις χώρες όπου βρίσκονται τα κεφάλαια, που συνήθως είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο συμβιβασμό που προτείνεται αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι περίεργο. Αναφέρεται ότι αν τα κεφάλαια διαχειρίζονται από κάπου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει ότι το κεφάλαιο συμμορφώνονται με κάποια κριτήρια. Όμως, αν η διαχείριση γίνεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες, δεν του ζητάει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δίνουμε κίνητρα στους διαχειριστές των κεφαλαίων να φύγουν από το City του Λονδίνου και να πάνε στη Νέα Υόρκη. Αυτό θέλουμε. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να πούμε ότι ακόμη και αν ο διαχειριστής βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάζει αν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις στη χώρα όπου βρίσκεται το κεφάλαιο. Όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο. Είχε προτείνει τρία χρόνια η Κομισιόν, εσείς προτείνετε τρία συν δύο, πέντε δηλαδή. Το πολιτικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε όμως δεν μπορεί να είναι περιμένουμε πέντε χρόνια και μετά κάνουμε κάτι. Αν δεν γίνει τίποτα τα δύο πρώτα χρόνια και δεν γίνει και τίποτα μετά μέχρι να τελειάσουν τα πέντε χρόνια καταλήγουμε σε ένα αδιέξοδο στο τέλος που δεν βοηθάει κανέναν γιατί καθυστέρησε γενικά η διαδικασία. Πρέπει να έχουμε μια μεταβατική περίοδο, όμως να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που να διασφαλίζουν ότι όντως θα υπάρξει μετάβαση, θα έχει ξεκινήσει μετάβαση και ότι θα μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετάβαση. Άλλο θέμα ενεργητικό και παθητικό marketing. Στην ε, συμβιβαστική λύση που προτείνεις υπάρχει μια παράγραφος που μας, που μας επιτρέπει να λύσουμε το θέμα γιατί αναφέρεται ότι αν διαχειρίζεται αν κεφάλαιο το διαχειρίζονται από εκτός, από χώρα όπου δεν υπάρχει ισοτιμία, τότε αναφέρεται στην παράγραφο αυτή ότι ο επενδυτής δεν έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να παραμείνει στον τελικό συμβιβασμό γιατί διαφορετικά ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας και ό,τι και να κάνουμε στην οδηγία, αν δώσουμε τη δυνατότητα στους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν ε, την οδηγία για το παθητικό μάρκετινγκ για να αγοράζουν κεφάλαια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το μόνο που κάνουμε είναι να δημιουργούμε προβλήματα για τους φίλους μας στο City του Λονδίνου, χωρίς να βοηθούμε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ, Σαΐτ. Θες να μιλήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να, να μην πω συγχα... συγχαρητήρια αλλά εκτιμώ τη δουλειά που έκανε ο Ζαν Πολ μέχρι τώρα προσπαθώντας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξει κάποιες συμβαστικές αρχές και τροπολογίες για να συζητήσουμε ενδεχομένω. Ο χρόνος που χρειάστηκε έχοντας να διαβάσει τόσες τροπολογίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δείχνει ότι είναι πολύ ικανός και αυτή είναι μια φιλοδοξία μου, δική μου, να μπορώ να χωνεύσω 1669 τροπολογίες του σύντομα και να καταλήξω συμβιβασμού. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τις συνεδρίες των σκιωδών συγκητών τη Δευτέρα ήταν ότι εκτιμήθηκαν οι διάφορες θέσεις. Αν δείτε τις θέσεις στην Επιτροπή υπάρχουν δύο άκρα και πρέπει να βρούμε συμβιβασμό μεταξύ των δύο. Ένα από τα άκρα είναι ότι η μία τοποθέτηση ακραία είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κάτι παρόμοιο με τη ΣΥΠΑ ή τη Σιγκαπούρη. Να μην προχωρούμε πιο πέρα. Δούμε την καταχώρηση, η αποκάλυψη στοιχείων, κάποια υποβολή αναφορά στο συστημικό κίνδυνο. Και αυτή θα ήταν η πρώτερη θέση μου αλλά όλοι μετακινηθήκαμε στη συζήτηση. Το είπε και ο εισηγητή στην προηγούμενη αλλαγή απόψεων και αυτό μετακινήθηκε. Άλλη ακραία θέση. Υπερβολικά προστατευτική. Απαγόρευση σε πόρου Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ευρωπαϊκά, να καταστρέψουν την οικονομία των ίσων Καϊμάν. 57% είναι οι υπηρεσίε των ίσων Καϊμάν, επειδή δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και να μειώσουμε τι συντάξει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιε αυτέ τι αντιλήψει. Υπάρχει αντίληψη ότι τα ταμεία επενδύουν πολλά χρήματα στα hedge funds ένα μικρό ποσοστό πηγαίνει στα hedge funds για να έχουν κέρδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να δούμε ποιο είναι επαγγελματία πελάτη και επαγγελματία επενδυτή και ο λιανικό επενδυτή και τι διαφορέ που υπάρχουν λόγω τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Προστασία του τομέα τη λιανική. Κάποιο μου είπε ότι είναι ο μεγαλύτερο ελέφαντα στο μικρό νησί. Τα νησιά Κέιμαν ε, είναι κίνδυνος οι νήσοι Κέιμαν έχουν περίπλοκη νομοθεσία για τα οικονομικά, περισσότερο από ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ φορολογική ουδετερότητα και φορολογικού παραδείσου. Τώρα για τις συμβιβαστικέ λύσεις που προτάθηκαν. Αναφέρονται σε κάποιες αρχές της ισοδυναμίας, αντιστοιχία. Ε, δίνεται πολλή εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άποψή μου. Θέλω να εξετάσω λεπτομερέστερα τι προτάσει για την αντιστοιχεία ισοδυναμία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλει κανονισμό για συνετή διαχείριση. Οι, Ευρω... Αμερικανοί θα το δεχτούν αυτό. Θα εστιαστούν ε, στι τράπεζε στο θέμα του περιθωρίου και του μεσάζοντε. Θα μπορούσε να μα διαφωτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως θα πρέπει να δίνεται χαρακτηρισμός ευρωπαϊκός για ευρωπαϊκούς ε, τα, πόρους, ευρωπαϊκά ταμεία με ευρωπαϊκή ετικέτα, ευρωπαϊκό τίτλο. Χαιρόμαστε όταν χρησιμοποιούμε αυτή την ετικέτα, αν θέλετε, αυτό το χαρακτηρισμό στη, στην Ασία, παρόλο που δεν ζητούμε αντιστοιχεία στις ΗΠΑ. Τι πρέπει να εξετάσουμε. Έχει κανείς ένα ταμείο ή διαχειριστή πόρων που δεν πληρεί τα κριτήρια ισοδυναμίας εκεί που υπάρχουν διάφορα σχήματα εθνικά ιδιωτικών επενδύσεων σε επιτραπεί να συνεχίσουν. Και θα πρέπει η Εθνική Αρχή να αναφέρεται στην ΕΣΜΑ για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί θέλουμε να μειώσουμε τα κέρδη των εξωτικών ταμείων. Λόγω προστατευτισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. λόγω διακριτική μεταχείρισης κατά των μικρών νησιών της Καραϊβική. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε. Συμφωνώ με τον Wolf όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή πρέπει να εξεταστεί. Συμφωνώ με τον Βολφ, με τον Ρόμπερτ, τον Ρόμπερ Γκέμπελς. Και κάτι άλλο. Θα πρέπει οριζόντια να υπάρχει πρόθεση στο παιδί αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν διαφορές εκεί όσον αφορά το short selling. Ας το εξετάσουμε οριζοντίως. Εκτιμώ τη θέση του συγγητού όσον αφορά τη μόχλευση κατανοεί την ανάγκη να εξεταστεί κατά περίπτωση το φαινόμενο της μόχλευσης. Τα, οι διάφορες τάξεις στοιχείων ενεργητικών, οι αρμόδιες αρχές όπως η ΕΣΜΑ να κατευθύνει τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Όσον αφορά τις προτάσεις του για τις αμοιβέ. Σαΐντ, Πιο σιγά σε παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρο. Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, ναι, θα πάω πιο αργά. Προσπαθούσα να βιαστώ. Ίσως να μου δώσετε άλλο ένα πεντάλεπτο τουλάχιστον. Τελευταίο σημείο, οι αμοιβέ. Είναι καλό το ότι εκτιμούμε τις διαφορές που υπάρχουν για εκείνους που χειρίζονται τα ταμεία και τις τράπεζες, ότι υπάρχει διαφορά. Είναι σημαντικό για μας. Εκεί που οι τραπεζίτες αμοιβόταν ακόμα και για κακές επιδόσεις. Υπάρχουν διαφορετικές δομές όσον αφορά τις αμοιβέ στη διαχείριση των πόρων και των ταμείων. Εκτιμώ τα όσα έκανε ο σχετικά. Έχουμε και τις δύο ακραίε θέσει. άρα υπάρχει περιθώριο λιγμών μεταξύ των δύο. Και σίγουρα με τι δέσμε προσπάθειες θα πετύχουμε τον αναγκαίο συμβιβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλουτ, επόμενος σκιώδης. Ο κύριος Κλουτ, ευχαριστώ. Ζαν Πολ δεν ήταν κάποιο που ζηλεύαμε για την πολλή δουλειά που συνεπάγεται αυτό. Αυτό το υπενυχτήκαμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ για το έργο που έκανε. Υπάρχουν κάποια επιμέρου σημεία που υπό το πρίσμα το δικό μου θα ήθελα να αναφέρω. Υπό τις τροπολογίες υπήρξε μια σειρά τροπολογιών που πρότειναν όχι μόνο το IFM να αναφέρεται αλλά το ίδιο το Ταμείο εδώ θα ήθελα από σένα, Ζαν Πολ, να ακούσω ποιο είναι το σχόλιο σου, πώς αντιμετωπίζεις εσύ το θέμα αυτό, τι προτείνεις μετά από τα όσα προτάθηκαν από εμά. Ένα άλλο θέμα, το θέμα των μικρών, μικρότερων ταμείων. Το γνωρίζω αυτό το επιχείρημα. Έχει προηγούμενα αναφερθεί, αλλά και τώρα Τίθεται εδώ βέβαια το ερώτημα αν είναι σκόπιμο αυτό να γίνει ή όχι. Ξέρω τα επιχειρήματα αυτών που κατέθεσαν προτάσεις τουλάχιστον από την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Λένε εφόσον σε, εθνικ, σε επίπεδο κράτους μέλους πρέπει να υπάρχει υψηλή, υψηλό επίπεδο ρύθμισης. Λογικό αυτό, αλλά να ρωτήσει κανείς αν σε εθνικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει επιπλέον ρύθμιση, τότε αυτό είναι διπλό επικάλυψη. Δεν είναι το καλύτερο για να καταλήξουμε σε ρύθμιση στο ευρωπαϊκό επίπεδο, να έχουμε διπλές ρυθμίσεις. Αυτό είναι που θα ήθελα να τοποθετηθεί ο κ. Γκοζές γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η διπλή, ας το πω έτσι, υπόθεση ρύθμισης. Έχει νόημα να γίνεται αυτό ή όχι, αυτό είναι ερώτημα. Τώρα, ένα άλλο σημείο και πριν από αρκετό χρόνο το είχα αναφέρει. Η αριστερή, η Γκουε, προγραμματικά ζητάμε να υπάρξει απαγόρευση hedge funds, hedge funds και private equities. Φυσικά δεν μπορεί να τύχει πλειοψηφική έγκριση αυτό, το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό για μας ε, η ρύθμιση για την μόχλευση έχει σημαντικό ρόλο. Θέλω να υποστηρίξω αυτό το οποίο είπατε εσείς πιο πριν ότι οι τράπεζες διαδραματίζουν εδώ ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και τουλάχιστον στην Ομοσπονδιακή Γερμανία υπάρχουν αρκετοί που κατά το τελευταίο διάστημα κατέθεσαν αυτή την άποψη στη δημόσια συζήτηση ότι πιθανόν εδώ πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση ή να τραβηχτεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ ταμείων και τραπεζών Δηλαδή, ο τομέα των επαγγελματικών τραπεζικών δραστηριοτήτων πρέπει να διαχωρίζεται από τον άλλο. Πώ θα γίνει αυτό, υπάρχουν αρκετέ προτάσει. Αν θα ήταν δυνατό αυτό να γίνει, θα το χαιρέτιζα. Υπό αυτό το πρίσμα να υπάρξει κάποια ρύθμιση που θα μπορούσε να ενταχθεί. Όπω ε, το υπενηχθήκατε. Το βρίσκω πραγματικά αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερα σκόπιμο. Προστασία των συνταξιούχων η πείρα στην Αμερικανική κρίση κατέδειξε πόσο οι ασφαλίσεις συντάξεων συνταξιοδότησης μπορούν να υπονομευθούν και να καταστραφούν. Πρέπει να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που εργάστηκαν όλη τους τη ζωή για να πάρουν μια σύνταξη να δουν να χάνονται τα χρήματά τους ξαφνικά. Τα χρήματα στα οποία έλπιζαν ότι θα πάρουν και στα τα οποία υπολόγισαν ξαφνικά να εξανεμιστούν για τις αμοιβέ πρέπει να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπα. Πρέπει να είναι σαφές ότι θα υπάρχει μια αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης που θα αποκομίζει κανείς βλέποντας αυτές τις ρυθμίσεις. Τελευταία παρατήρηση, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, θέλω να το υπενθυμίσω αυτό γιατί το βρίσκω σημαντικό που στοχεύουν στην ε, αγορά κάποιων μημάτων ε, επιχειρήσεων μέσω των ταμείων ε, να υπάρχει και ενημέρωση σε σχέση με τους εργαζόμενους. Είναι καθήκον αυτό να γίνεται. Δεν πρέπει να το αγνοήσουμε και να μεληθεί. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία τώρα που σε σχέση με τον Ζαν Πολ έχει από πλευρά ε, συμβιβασμών τονιστεί ιδιαίτερα. Αισθάνομαι όμως ιδιαίτερη υποχρέωση να μην ξεχάσουμε αυτή την πτυχή για τους εργαζόμενους. Ε, να βρεθεί μια σαφής ρύθμιση οι εργαζόμενοι οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους να ενημερώνονται, να πληροφορούνται όταν τέτοιου είδους ε, ταμεία δρούν αυτόν τον τρόπο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Προχωράμε. Θα πρέπει όμως να είστε πιο σύντομοι από τους σκιώδεις εισηγητής. Ξεκινάμε με την Άστριτ Λούλινγκ. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω όμως κάτι όσον αφορά το Συμβούλιο και την τελική εξέταση θα μπορούσαμε βεβαίως να ανησυχούμε για αυτή την έκθεση που δεν ξεκινάει τίποτα καλό και να διαπιστώσουμε ότι το Συμβούλιο θα καταλήξει σε απόφαση μετά από πολλές διαπραγματεύσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως το Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να θέτει το πύχη πολύ ψηλά γιατί οι διαπραγματεύσεις κρατούν πολύ και ευτυχώς συμφωνεί και ο εισηγητής ότι δεν είναι εύκολο να καταλήξει σε καλή απόφαση το Συμβούλιο γιατί υπάρχουν πολλά συμφέροντα και άρα το έργο μας εδώ στο Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό γιατί μόνο εμείς μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα και επίσης ικανοποιητικό και συνεκτικό. Πιστεύω ότι θα κερδίσει πολλά η Επιτροπή μας λοιπόν αν καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσον αφορά τους συμβιβασμούς που προτείνονται μετά από τις πρώτες διαπραγματεύσεις. Κάποια σχόλια. Καταρχάς όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Ε, μένω ικανοποιημένη από το γεγονός ότι κινούμαστε προς την εσωτερική αγορά. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Κλίντς Συμφωνώ αυτή τη φορά με την ΚΟΕ όσον αφορά την κατάτμιση της εσωτερικής αγοράς. Θεωρώ ότι τα εθνικά και διεθνή κεφάλαια θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση. Και εγώ τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαι, έχοντας ακούσει και τον κύριο Γκέμπελ στο συμπρατηριότη μου. Όσον αφορά τώρα τα κατόφλια, νομίζω ότι είναι λογικό να μην έχουμε κατόφλια. Πρέπει να ελέγχονται όλα τα κεφάλαια, αλλά αναλογικά. Έχοντας ακούσει τον εισηγητή όμως πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια λογική λύση στο πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα τα εναλλακτικά κεφάλαια σε τρίτες χώρες. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει επιληθεί ακόμη ικανοποιητικά. Αν κινηθούμε προς ένα σύστημα ισοτιμιών θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους κανόνες που θα επιλέξουμε για το παιχνίδι. με καθησύχασαν κάποια πράγματα που άκουσα, αλλά να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είδα λομπίστες από τα νησιά Κάιμαν και μου είπαν ότι οι προδιαγραφές τους είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο. Εντάξει. τότε τους είπα ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με ένα πρόβλημα μόνο με έπεισαν ότι θέλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις προδιαγραφές που θα απαιτήσουμε. Με αυτό συμφωνώ. Πρέπει από την αρχή να θέσουμε σαφείς κανόνες. και όχι να περιμένουμε να περάσει κάποιος χρόνος πριν να διαπιστώσουμε αν υπάρχει ισοτιμία ή όχι. Αυτό είναι σημαντικό για εμένα. Πρέπει οι τρίτες χώρες να γνωρίζουν εκ των προτέρων ακριβώς τι εννοούμε. Ένα δεύτερο θέμα. Όσον αφορά τα εθνικά συστήματα τα εθνικά private equities. Και εκεί νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λογική λύση. Να πω πάντως ότι το σύστημα ισοτιμιών με βάση ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο έχει πολύ λίγες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο, άρα ίσως θα έπρεπε να βρούμε ένα μηχανισμό λιγότερο φιλόδοξο, λιγότερο πολύπλοκο. Και κάτι τελευταίο για τους καταθέτες. Είχα πει και πριν ότι πρέπει να αποσαφηνίσουμε περισσότερο τις ευθύνες των καταθετών γνωρίζοντας τα προβλήματα που είχαν υπάρξει, όμως να μην πάμε και υπερβολικά μακριά για να μην καταλήξουμε σε ένα σύστημα αναποτελεσματικό και δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για συναλλαγές οι οποίες, τις οποίες μάλλον δεν μπορούν να ελέγξουν. Επίσης, στα πλαίσια του συμβιβασμού θα έπρεπε να δούμε τα θέματα τόσο της διασφάλισης ε, των ε, στοιχείων αλλά ολοκληρώνοντας να πω ότι χαίρομαι πολύ για τις εξελίξεις δεν ξέρω, δεν θέλω να σε συγχαίρω και πολύ Ζαν γιατί ίσως το παρανοήσουν κάποιοι Ευχαριστώ. Να διαβάσω ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο και μετά να δούμε ποιοι θα χωρέσουν. Annika Jury, Udo Bullman, Corinne Wortman Cool, myself, the Commission if they're extremely lucky, and then the rapporteur again. So, Peter, it's you. Thank you very much, and thanks again to Jean-Paul. Peter, Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Ζαν Πολ για το ότι έχει κάνει μέχρι στιγμής, ειδικά όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Είναι χρήσιμο αυτό που έχεις κάνει και εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να εξαιρούμε, πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε. Υπάρχει αυτή η διαστρεβλωμένη άποψη ότι λόγω μεγέθους κάποια δεν σημαίνουν κάτι. Δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό το είχαμε ακούσει και για τις τράπεζες όμως. Επίσης συμφωνώ που μιλάς για αναλογικότητα. Είναι πολύ θεμελιώδες ζήτημα και συμφωνώ μαζί σου. Έχοντας συναντηθεί και με Γάλλους τραπεζίτες, συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε τους κανόνες και να τους δίνουμε τη δυνατότητα να μπορούν να αντιδρούν με τον κατάλληλο τρόπο. Άρα τίθεται και θέμα διαλειτουργικότητας όσον αφορά τις τρίτες χώρες και το short selling. Καταθέσει σε τρίτες χώρες και short selling. Τα έχουν ήδη πει κάποιοι, αλλά είναι σημαντικά. Χτες ε, συναντήθηκα με έναν Άγγλο που ζει στην Αμερική και κατασκευάζει φωτοβολταϊκές πίνακες. Πήγε στην Αμερική και του έδωσαν 500 εκατομμύρια για να επενδύσει. Έτσι απλά. Εντάξει, όχι έτσι απλά, αλλά παρόλα αυτά εντυπωσιακά απλά. Και ξέρετε, έχει ηγετική θέση η Ευρώπη σε αυτή τη τεχνολογία, ειδικά η Γερμανία. Όμως η επένδυση σε αυτό το πράγμα θα γίνει στην Αμερική γιατί είναι πιο εύκολο. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι αυτά τα ιδιωτικά κεφάλαια έρχονται συχνά γιατί είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν αλλού εκτός Ευρώπης και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Δεν μπορούμε να στριμώξουμε τον ε, καπιταλισμό στη γωνία και να πούμε ότι δεν θα λειτουργείτε καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε και γνωρίζω ότι είστε ρεαλιστής, άρα θα το έχετε υπόψη σας. Τώρα όσον αφορά τις τρίτες χώρες και τη δυνατότητα συμμετοχή τους στη δραστηριότητα στο μέλλον. Εγώ ανησυχώ πολύ όταν μιλάμε για τρία με πέντε χρόνια και μιλάμε για ισοτιμίες. Έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα των ισοτιμιών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απαγαρεύουμε προϊόντα ή διαχειριστές γιατί εμείς έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένο επίπεδο για τις αγορές μας Κοιτάξτε, το θέμα θα έπρεπε να είναι τα οι διεθνείς προϋποθέσεις, οι παγκόσμιες προϋποθέσεις, όχι μόνο οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ίσως δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη σύγκληση, αλλά πρέπει να έχουμε μια κοινή πορεία όσον αφορά το πώς αυτές οι προδιαγραφές προστατεύουν τους επενδυτές και λειτουργούν καλά τα καθεστώτα. Άρα πρέπει να έχουμε ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά την ισοτιμία, γιατί αν δεν το κάνουμε θα είναι σαν να απαγορεύουμε την πρόσβαση σε όλους τους εξωτερικούς επενδυτές. Για παράδειγμα αυτούς που επενδύσανε 500 εκατομμύρια για τα φωτοβολταϊκά. Και Είπε η κυρία Λούλινγκ ότι συναντήθηκε με τραβαζίτες. Χαίρομαι γι' αυτό. Όμως, κοιτάξτε, στο... με την υπόθεση Μέιντοφ χάθηκε 1,6 δισεκατομμύριο παρά την ρυθμιστική διαδικασία παρά τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν άλλου. Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καλές προδιαγραφές για την προστασία των επενδυτών πρέπει να ασχοληθούμε τους διαχειριστές των κεφαλαίων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάχρηση. Και λυπάμαι, Ζαν Πολ, που δεν τον λαμβάνεις υπόψη του. Μας λες ότι θες να προστατεύσεις τους επενδυτές. Τι θα κάνουμε όμως με τους Γάλλους επενδυτές που έχασαν λεφτά λόγω του Μέιντοφ. Ας τους λάβουμε υπόψη μας για να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. Και όσον αφορά το short selling, όντως θα έπρεπε να είναι οριζόντιο θέμα, γιατί με ανησυχεί ο ορισμός σου. Λες ε, οποιαδήποτε καταθρηστική και χειραγωγική διαδικασία αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην οδηγία για τις αγορές. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια καλή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σημεία είναι τα σημεία κίνησης, θα έλεγα, για αυτή τη συζήτηση. Ένα, ότι όλοι πρέπει να ευγνωμονούμε το Ζαν Πολ που δούλεψε έτσι. Όσο πιο πολύ μελετώ τις τροπολογίες, πρέπει αυτό να το τονίσουμε τόσο το περισσότερο Πραγματικά εδώ υπάρχει και κίνδυνος να σου απονεμηθεί και νομπέλ. Είναι τρομερή δουλειά που έκανες, πρέπει να το ομολογήσουμε. Το δεύτερο σημείο εκκίνησης. Αυτό είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό που, που κάνουμε εμείς εδώ συνεισφέρει στις ε, χρηματοοικονομικές αγορές της Ευρώπης ότι συνάδει με τους στόχους που έχουμε για παράδειγμα για την Ατζέντα 2020. Όταν κάμια φορά παρακολουθώ τη συζήτηση για τα εναλλακτικά ταμεία επενδύσεων Alternative Investment Funds πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να συνεισφέρουν αυτές οι επενδύσεις στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αυτή είναι η σωστή ισορροπία που πρέπει να διασφαλίσουμε εδώ. Τώρα, όσον αφορά το φάσμα, το εύρος αυτής, τη της προσπάθειας, εκτιμώ αυτά τα οποία συντάχθηκαν για τις βιομηχανικές εταιρείες ε, μερισμάτων, όμως θα πρέπει να το βελτιώσουμε στα σκεπτικά, στις αιτιολογικές σκέψεις ε, σε σχέση με αυτή την οδηγία να αποσαφηνίσουμε ότι οι εταιρείε που ασχολούνται με επενδύσεις, ε, βιομηχανικές επενδύσεις δεν θα εντάσσονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεύτερον όσον αφορά τρίτες χώρες. Από ό,τι κατάλαβα ο εισηγητής δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη δουλειά σε σχέση με τον συμβιβασμό, συμβαστική λύση που προτείνεται γι' αυτό και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα ως τελική έκβαση, ως κοινό παρονόμαστη <clears throat> θα πρέπει εμείς όσον αφορά τους, τις ΙΠΑ ή τις ασιατικές χώρες δεν θέλουμε να έχουμε δεσπόζοντα ρόλο εκείνοι να ακολουθήσουν εμάς πρέπει να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή κανονισμών, διατάξεων κτλ. Διότι οτιδήποτε και αν θεωρούμε ένα μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου κόσμου θα παραμείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα είναι υποφελές αν εμείς συνεχίσουμε εμείς να θέτουμε τον εαυτό μας εκτός αυτών που είναι σημαντικά όχι μόνο για εκείνους που ε, αποταμιεύουν για τις συντάξεις τους αλλά χρειαζόμαστε και μια σωστή ρύθμιση σε σχέση με τις τρίτες χώρες και να τονιστεί σε σχέση με το Συμβούλιο η ανάγκη εμείς ως Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη ε, διαδικασία, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα επανέλθω φυσικά επίσης και στη συζήτηση που έγινε όσον αφορά τα κατόφλια και την αναλογικότητα. Τώρα στις συμβαστικές προτάσεις έχουμε ένα συνδυασμό κατοφλίων με το άλλο θέμα. Είναι ένα τρόπο με τον οποίο αποσαφηνίζουμε πώ θα πρέπει να προσαρμοστεί η αρχή τη αναλογικότητα και θα λειτουργήσει. Όμω θα πρέπει το επίπεδο κατοφλίων να επικεντρώνεται σε σχέση με τα κατόφλια όπου εμφανίζονται συστημικοί κίνδυνοι. Θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή, το επίπεδο των κατοφλίων αυτών. Αυτό σίγουρα μπορούμε να το συνεχίσουμε στη συζήτησή μα τι επόμενε εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ σε σχέση με το βραβείο Νόμπελ δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Ίσως όμως μπορείτε να ανακηρυχθείτε Ευρωβουλευτής της χρονιάς. Όμως θα ήθελα να συγχαρώ. Νομίζω ότι πραγματικά κάνετε πάρα πολύ καλή, εξαιρετική δουλειά. Είναι η πεμπτουσία αυτό του να είναι κάποιος ευρωβουλευτής, να πετυχαίνει συμβιβασμούς και με ένα ευγενικό και με τριόφρον πνεύμα. έτσι να κερδίζουμε κάποια πράγματα ε, από, απεμπορώντας κάποια άλλα. Όμως είσαστε εξαιρετικό σε αυτό το εγχείρημα. Υπενθυμίζοντας αυτό που είπε ο κύριος Στρόσκαν, ότι δεν θα πρέπει μόνο να επικεντρωνόμαστε σε ρυθμίσεις και διατάξεις. Θα πρέπει στην εποπτεία, στην επιτήρηση να επικεντρωνόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποιοι από εσά πιστεύετε ότι μπορούν να ρυθμιστούν σχεδόν τα πάντα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό και το γνωρίζετε. Εγώ συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είχαμε ένα σωστό πλαίσιο ισορροπίας, ισορροπιών όσον αφορά τις διατάξεις. Αλλά μπορούμε να αναφέρουμε και το παράθυμα του Επιτρόπου Μπαρνιέ. Σε σχέση με τα όσα ανέφερε, υπενθύμισε ότι δεν ήταν τα hedge funds που προκάλεσαν την κρίση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε. Τι είπες Ρομπέρ, δεν το άκουσα εκτός μικροφώνου. Ναι, φυσικά μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση, να κάνουμε συζήτηση. Αλλά και σε κάποιους τομείς πιστεύετε κάποιοι από εσά ότι η, από πλευρά επιτρόπου θα ήθελαν όλα, όλα θα ήθελε να τα ρυθμίσει, αλλά έκανε αυτή την παρατήρηση, το υπενθυμίζω. Σύντομα σχόλια. Το θέμα τρίτο, τρίτης χώρας, τρίτων χωρών έχει ζωτική σημασία. Δεν χρειάζεται το επαναλάβω. Ουσιαστικά τον συμβιβασμό του Δεκεμβρίου της Σουηδικής Προεδρίας που ήταν αρκετά καλός πρέπει να πω. Όμως κατανοώ ότι ξεπεράσαμε ήδη αυτή τη φάση πια. Είναι πίσω μας πια και βρισκόμαστε εμείς αλλού. Φυσικά για τις συζητήσεις που ανέφερε ο Βολφ Κλίντς. Ουσιαστικά Βολφ η απόρριψη της τροπολογίας δεν ήταν εκείνος που πρότεινε αυτή την τροπολογία. Εγώ ήμουν και ο Βολφ που την προτείναμε. Βρισκόμαστε στο ίδιο σκάφο εμεί, αλλά το ξέχασε ο Βόλφ αυτό. Δεν πειράζει. Με κάθε μετριοπαθία αν λέω αυτό. Το άλλο είναι το θέμα του short selling. Και εκεί πάλι σήμερα το πρωί ήταν εξαιρετική η εκδήλωση. Αν ακούσατε τον Στρός Καν και τον κύριο Ντράγκη. Αυτό το θέμα για την Ελλάδα, για την... και όλα αυτά τα συναφή είπαν, προσέξτε, πρέπει να υπάρχει αξιοπρεπής, ε, αξιοπρεπές πλαίσιο επιχειρημάτων, επιχειρημάτων εδώ και υπάρχουν αρκετές επιπτώσεις ε. εδώ οριζόντια πρέπει να το δούμε. Έχουμε την περίπτωση του short selling στη χώρα μου. Δεν τα πάμε και τόσο αρνητικά, έτσι. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Δεν πάμε τόσο άσχημα λοιπόν, έτσι μπορούμε νομίζω και μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αλλά εγκάρσια, οριζόντια πρέπει να το δούμε και να, να δρούμε. Ολοκληρώνοντας κάποια σχόλια από πλευρά ε, κάποιου που παρακολούθησε το έργο αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πάνω από ε, δέκα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και αυτός ο άνθρωπος τι είπε, είπε ότι κάποτε στη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή πιστεύαμε και εσείς πιστεύατε ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας είναι ένα αξιόλογο τμήμα, μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς. Και αν αυτό αμφισβητηθεί, ε, αυτό που κάνουμε τότε εδώ δεν είναι ένα αξιόλογο τμήμα για τη δουλειά του χρηματοοικονομικού τομέα. Τουλάχιστον θα έπρεπε να ακούσουμε αυτά τα επιχειρήματα. Εσείς το κάνετε αυτό κύριε Γκοζές και βασιζόμαστε στη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος σας ευχαριστώ. Λούντβιξον παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ. Το Συμβούλιο αυτό το θέμα ήδη πριν από μια εβδομάδα το εξέτασε. Αν θέλουμε επικοδομητικά να καταλήξουμε στην εξέβρεση ενός συμβιβασμού και να καταλήξουμε σε ένα θετικό τελικό αποτέλεσμα ως έκβαση, τότε θα πρέπει να δράσουμε, να κινητοποιηθούμε ε, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις. Εναλλακτικές ε, ε, επενδυτικές δυνατότητες ως ταμεία είναι σημαντικό στοιχείο. Εδώ υπάρχουν θετικές προοπτικές όσον αφορά τις θετικές προθέσεις του εισηγητή. Όσον αφορά το θέμα της τρίτης χώρας. Είναι αποδεκτή αυτή η λύση θα έλεγα. Αυτή η λύση αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Μεταβατική περίοδος, ένα διαβατήριο, η η το Ταμείο Τρίτης Χώρας, πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ με αυτό το πάσο, με σαφή κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούνται ώστε να μπορούν να, να είναι αναγνωρίσιμα και να είναι αποδεκτά. Μια θετική και ελαστική συνεργασία και η τήρηση των κριτηρίων φυσικά που πρέπει πάντα να υλοποιούνται και να συμμορφωνόμαστε με αυτά. Τώρα, τούτων λεχθέντων. Θα έλεγα ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο κάποια προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν. Στην Ευρώπη σε σχέση με αυτό δεν πρέπει να οικοδομήσουμε σε σαθρά θεμέλια. Δεν μπορούμε υποχρεωτικά να προσανατολιστούμε με ε, γνώμονα το αμερικανικό πρότυπο, ακόμα και αν καμιά φορά φαίνεται ότι έχει κάποια προτερήματα. Και όσον αφορά και τις private equities, φαίνεται να είναι καλή λύση. Είναι λοιπόν σημαντικό, σίγουρα, σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπορούν να δίνουν πληροφορίες που είναι σημαντικές και πρέπει να ε, συλλέγονται. Αυτή η ίδια υποχρέωση πληροφόρησης και ενημέρωσης ισχύει για όλες τις ε, επιχειρήσεις, για όλες τις εταιρείες. Είναι κάτι το οποίο έχει καθορίσει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, όρο, προϋπόθεση που πρέπει να υλοποιείται. Πρέπει απαιτήσει πληροφόρησης να τίθενται στο μέγιστο, υψηλότερο επίπεδο από πλευράς των επιχειρήσεων, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες πληροφόρησης. Ταυτόχρονα φαίνεται να έχουμε προσεγγίσει αρκετά μια καλή λύση, πρόσβαση, προσπερασιμότητα σε κεφάλαια και κεφαλαιοχικές αγορές. Πολύ σημαντικό για αυτό το τμήμα. Ευχαριστώ. Άνεκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Κοζές, για την έξοχη δουλειά που έκανε, υπέροχη δουλειά του και θα ήθελα να πω ότι είμαι αισιόδοξη όσον αφορά την επαναφορά των κατοφλίων. Ήταν στην πρώτη εκδοχή της προτάσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα σαν αποτέλεσμα των συμβαστικών τροπολογιών νομίζω ότι τα κατόφλια επανέρχονται. Νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα κατά των κατοφλίων. Θα ήθελα όμω να σε πιστήσω την προσοχή επί της αναγκαιότητα αυτών. Η αυθαίρετη διαμεσολάβηση είναι ένα επιχείρημα αν δεν υπάρχουν τα κατόφλια και θέλει κανείς να ρυθμίσει όλα τα ταμεία. Ακόμα και μεσαίου μεγέθου ταμεία αντί αυτή περιπτώση θα πάνε σε τρίτες χώρες λόγω του διοικητικού άχθους και τότε προϊόντα από αυτά τα ταμεία θα βρουν το δρόμο τους προς την ευρωπαϊκή αγορά μέσω παθητικού μάρκετινγκ. Ε. Και νομίζω ότι διεφάνει από τη συζήτηση ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις, τους μικρότερους φορείς της οικονομίας μας και δεν θέλουμε να αυξήσουμε το γραφειοκρατικό άχθος που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Το άλλο επιχείρημα είναι το εξή. Αν αυτά τα ταμεία αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα παραμείνει ένα κενό στο προπολογισμό μας. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το ανεχθούμε τώρα, να τα αντέξουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ούτε. Ούτε Μπούλμαν, πολλά πράγματα αναφέρθηκαν. Δεν ξέρω αν το Συμβούλιο κάνει, ήθελε να κάνει χάρη στο Ζαν Πολ με την απόφαση που έλαβε. De facto όμως αυτό έκανε. Το έκανε χάρη, όποια πρόθεση και αν είχε. Πιστεύω ότι ο Ζαν Πολ με αυτόν τον τρόπο, με τον Ζαν Πολ εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή, για άλλη μια φορά ενδυναμωμένοι περνάμε στο προσκήνιο και καθόμαστε ως οδηγοί στη θέση οδηγού. Αναλαμβάνουμε τα ενία και έτσι για αυτούς τους συναδέλφους που σίγουρα με γνώση της ε, ουσίας ε, αλλά και με επιφυλάξεις ε, είπαν κάποια πράγματα ναι, αναφέρθηκε από πλευρά Όλε Σμιτ για παράδειγμα, έτσι, σήμερα το πρωί, ότι τα hedge funds δεν ήταν η πρωταρχική υπέτη τη οικονομική κρίση. Όμω δεν πρέπει να σμικρίνουμε το ρόλο του και να τα ωρεοποιούμε τα πράγματα και σε σχέση με την δράση μη ας το πω έτσι, εντάξει ταμείων και την ανεύθυνη πολιτική που ακολουθούν, έτσι οι ε, εμπριστές ε, επιταχύνουν το έργο τους ε, και υπάρχει ανεξέλεγκτη κατάσταση με βάση κάποιες κερδοσκοπικές δράσεις. Αυτά δεν εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο ευθύνη και υπευθυνότητα. Γι' αυτό γενικά να πω για το πλαίσιο και την ατμόσφαιρα, το κλίμα αυτής της συζήτησης, ναι, Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εμείς μπορούμε και πρέπει να αναλάβουμε νομοθετικό έργο. Ας μην έχουμε δισταγμούς. Πρέπει, μπορούμε να αναλάβουμε νομοθετικό έργο. Δεν χρειαζόμαστε να ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Έχουμε εντολή γι' αυτό από του πολίτε. Πρέπει θαραλέα να στραφούμε σε αυτή τη δουλειά του νομοθετικού έργου. Αυτό έκανε ο Ζαν Πολ. Έκανε σημαντικά βήματα και διαβήματα για το νομοθετικό έργο. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη ρύθμιση για τις τρίτες χώρες και να ρωτήσω σχετικά επαρκώς, επαρκούν αυτά τα οποία έχουν προβλεφθεί. Για παράδειγμα, φορολογικές ρυθμίσεις πάντα δίναμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα, διότι χωρίς λογικές και αποτελεσματικές ρυθμίσεις για τα θέματα φορολογίας και η ρύθμιση για τις τρίτες χώρες δεν μπορεί να δώσει αυτά τα οποία υπόσχεται. Θέλω να τονίσω λοιπόν εδώ για άλλη μια φορά ότι διαφορετικά από τον Wolf Klintz πιστεύω ότι για τα όρια μόχλευσης πρέπει εδώ να δώσουμε κάποια περαιτέρω πλαίσια. Τώρα, για την μοχλική ε, απόδοση σίγουρα είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά δεν είναι θέμα αυτορύθμισης. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι μπορεί με αυτορύθμιση να ρυθμίζεται. Δεν μπορούμε και στους αυτοκινητοδρόμους να λέμε στους οδηγούς εντάξει κύριοι, ρυθμίστε την ταχύτητά σας κατά το δοκούν εσείς οι ίδιοι μόνοι σας. Δεν γίνεται αυτό. Είναι κάτι που πρέπει ρυθμιστικά από πλευράς νόμου να γίνεται. Το ίδιο λοιπόν και πρέπει να γίνει κάτι με τα equity funds και να γίνει κάτι και το σημείο της ενημέρωσης και πληροφόρησης εργαζομένων όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πριν πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι πρέπει να είναι σεβαστό. Εδώ πρόκειται για τον περιορισμό της μοχλικής ε, απόδοσης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να δούμε στην περαιτέρω διαδικασία και ε, στους συμβιβασμούς. Πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Όταν αναφέρεται σε σχέση με τη συζήτηση σήμερα το πρωί κάτι, να λάβετε υπόψη ότι αναφέρθηκε από τους επαΐοντες επίσης ότι τα ταμεία κατά το ίμιση των βραχυπρόθεσμων ε, αυτών συναλλαγών είναι υπεύθυνα για αυτή την κατάσταση πραγμάτων. Και πρέπει να δούμε και τα θέματα των ακάλυπτων συναλλαγών. Δεν πρέπει να, κάνουμε, να, υπάρξουμε, να υπάρξουν εδώ συμβιβασμοί και να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με τα όσα έγιναν στα κράτη-μέλη. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι, να ρυθμίσουμε αυτό το πράγμα όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση εξαιτία των φόβων του Gordon Brown για τις ε, επόμενες εκλογές και γι' αυτό βρισκόμαστε τώρα στην ηγετική θέση εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τον Ζαν Πολ Γκοζές. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Γι' αυτό πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι δυνατό και είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτό να ευχαριστήσω τον Ζαν Πολ για το πολύ καλό έργο του και να σου δώσω και κάποια σχόλια που ελπίζω ότι θα σε καθοδηγήσουν περισσότερο στην οριστικοποίηση των συμβιβαστικών τροπολογιών. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, νομίζω ότι κινούμαστε προς τη στη κατεύθυνση. Αν και χρειάζονται περισσότερες αποσαφηνήσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες για το τι συμπεριλαμβάνεται και τι όχι. Νομίζω ότι σε κάποιες ε, περιοχές η ε, αναλογικότητα θα έπρεπε να εξεταστεί περισσότερο, παρόλο που σε πολλά σημεία συμπεριλαμβάνεται καλώς. Για παράδειγμα, οι εταιρείε οι οποίες βρίσκονται στο χρηματιστήριο πρέπει να συμμορφωθούν και με την οδηγία το άρθρο 30. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο, ίσως θα έπρεπε να το διαγράψουμε αυτό. Όσον αφορά τώρα τις τρίτες χώρες, είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το υπογραμμίσω να μείνουν ανοιχτές οι δυνατότητες για τους επαγγελματίες επενδυτές τρίτων χωρών οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να επενδύουν σε εναλλακτικά κεφάλαια με έδρα τρίτες χώρες. Οποιοςδήποτε περιορισμός, ειδικά όταν αφορά το private equity, είναι μάλλον περιττός, γιατί δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους κεφάλαια αποτελούν συστημικό κίνδυνο. Όσον αφορά τώρα την υποτίμηση και εκεί μπορώ να συμφωνήσω με τον ε, συμβιβασμό και το ίδιο και για τη μόχλευση, αν και νομίζω ότι ίσως χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων. Γι' αυτό να σας υπενθυμίσω για την πρόταση του Συμβουλίου, όπου οι εθνικές ελεγκτικές αρχές παίζουν ρόλο κλειδί στον καθορισμό των μέγιστων ορίων για την μόχλευση, καθώς επίσης και για την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου αυτών των κεφαλαίων. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να χρησιμοποιήσουμε την πρόταση του Συμβουλίου. Όσον αφορά τώρα τους ε, καταθέτες, Στην συμβιβαστική σας λύση προτείνεται να έχουμε ως τέτοιου είδους αποθετήρια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όμως, για παράδειγμα, στις κάτω χώρες έχουμε και άλλους οργανισμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να τους αποκλείσουμε. Αυτά είναι τα σχόλιά μου προς το παρόν. Καλή σας επιτυχία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε σε μια επιτυχή ψηφοφορία τον Απρίλιο. Ευχαριστώ. Και καταλήγουμε σε μένα από πλευράς Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν υποθεί πάντα πίστευα ότι ο στόχος μας ήταν να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να αντιμετωπίσουμε τους συστημικούς κινδύνους. Νομίζω ότι αυτή ήταν πάντα η προθέση μας. Γι' αυτό και δεν με ανησυχεί το γεγονός ότι έχει επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής πέρα από τους συστημικούς κινδύνους. Νομίζω ότι αυτό θέλαμε να κάνουμε με αυτή την έκθεση και στην προηγούμενη θητεία. Όσον αφορά τις τρίτες χώρες, θα θα ήθελα καλύτερη μεταχείριση όταν έχουμε τη μία πλευρά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε η μία πλευρά είναι το κεφάλαιο, είτε οι διαχειριστές του κεφαλαίου. Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδους έλεγχος των της κατάστασης. Και αυτό που φοβάμαι είναι αν ο διαχειριστής του κεφαλαίου είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως ε, εμποδιστεί να επενδύσει σε κάποια κεφάλαια. Στην πρώτη πρώτη ανταλλαγή απόψεων είχα αναφερθεί στις ε, μη αναπτυγμένες ε, ή αναπτυσσόμενες χώρες όπου δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ισοτιμία αλλά όπου ίσως να υπάρχουν ευκαιρίες επένδυσης. Δεν θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε την πόρτα σε αυτές. Θεωρώ ότι αν έχουμε διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε οι ελεγκτικέ αρχέ της Ευρωπαϊκής Ένωση θα μπορούσαν να έχουν κάποια δυνατότητα ελέγχου σε θέματα όπως η διαφοροποίηση και τα των επενδύσεων σε τρίτες χώρες. Υπάρχουν λοιπόν επιχειρήματα επ' αυτού. Όσον αφορά την ευθύνη για τα depositories, τα αποθετήρια, έχω πρόβλημα με την έκφραση force majeure, έκτακτης ανάγκης δηλαδή, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι όλοι πιέζουμε προς την ίδια κατεύθυνση εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα θα είναι απολύτως ε, υπεύθυνα για όλα τα αποθετήρια, τα καταθέτες, δεν νομίζω ότι εννοούμε κάτι τέτοιο, απλά χρειαζόμαστε να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση. Επίσης, να πω ότι μου άρεσε η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να αναθέσουμε σε τρίτους και να υπάρξει μία σύμβαση η οποία να αναφέρει σαφώς ποιος θα είναι ο υπεύθυνος. Να μην υπάρχει δηλαδή μια τέλειωτη αλυσίδα αναθέσεων και τελικά να μην γνωρίζουμε ποιος έχει την ευθύνη. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους περιορισμούς συμβοτικούς και κάτι τέτοιο θα με έβρισκε σύμφωνη, αν βρείτε την κατάλληλη διατύπωση. Όσον αφορά τη μόχλευση, ο Ούντο είπε ότι η μόχλευση είναι θέμα αυτορύθμισης. Συμφωνώ, αλλά επίσης μπορεί να είναι και ρυθμιστική παρέμβαση. Και υπάρχει περιθώριο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός των εθνικών κρατών για παρεμβάσεις. Οπότε γενικά μιλώντας θα έλεγα ότι η, ελεγκτική, η νέα ελεγκτική αρχή θα μπορούσε να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πότε θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν οι εθνικές ελεγκτικές αρχές. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία και είναι δύσκολο να θέσουμε απόλυτα περιοριστικούς κανόνες, σαφείς κανόνες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η άποψή μας. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε με τους άλλους ότι έχει προχωρήσει πολύ και θυμάμαι και την οδηγία για τις άμεσες πληρωμές και θυμάμαι ότι και τότε δεν μας έκανε καθόλου κακό η προετοιμασία στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Μας μένουν τρία-τέσσερα λεπτά. Ζαν Πολ, θες να ακούσεις την Επιτροπή, θες να μιλήσεις. Απλά να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα, αλλά ας περιμένουμε το τέλος της διαδικασίας για να δω αν τα ακουξίζω τα συγχαρητήρια. Να πω ότι στην πρώτη συνεδρίαση με τους ε, σκιώδεις εισηγητές είχαν προχωρήσει κάποια πράγματα και τώρα κάνουμε το ίδιο. Συνεχίζω το έργο μου και όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, αυτή η προετοιμασία μόνο καλό πράγμα μπορεί να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έληξε η συνεδρία μας εδώ, σχεδόν στην ώρα μας.